continuar con los Μπορούμε να περάσουμε στη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής μας και όπως γνωρίζετε είχαμε προηγούμενα μία συνάντηση με τον κύριο Γιουγνάν, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και τους συντονιστές. Είχαμε ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε και μερικές πριν από μερικέ ε, την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Υπουργό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα, πρώτον να του δώσουμε το λόγο. Θα ήθελα όμως ε, να τον καλωσορίσω σε αυτήν την Επιτροπή Αλία του Κοινοβουλίου για την παραδοσιακή παρουσίαση των προτεραιοτήτων της νέα Προεδρία του Συμβουλίου και μετά να σας δώσω φυσικά την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις ε, με τον κύριο Υπουργό. Σας είπα ήδη ότι η μεταρρύθμιση της κοινή ελεύθερης πολιτικής ε, τόσο ό,τι αφορά τον βασικό κανονισμό όπως και το ζήτημα των αγορών και σήμερα το πρωί εγκρίναμε την έκθεση αναφορικά με το σχετικό ταμείο και θα είναι και το πρώτο ζήτημα που θα συζητήσουμε με την Λιθουανική Προεδρία. Του αναφέραμε επίση κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα έλεγα ότι παραμένουν ένα σταθερό αίτημα της Επιτροπής μας για τα προγράμματα διαχείρισης τα οποία έχουν μπλοκαριστεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα επαναλάβουμε προς την Προεδρία, στην περίπτωση αυτή προς την Λιθουανική Προεδρία, να φροντίσει η υπόθεση αυτή να προχωρήσει, να αποδεσμευθεί. Επίση έχουμε και προσφυγικέ στο δικαστήριο, αλλά εμεί είμαστε πολιτικοί, πρέπει να βρίσκουμε πολιτικέ λύσει στα διάφορα προβλήματα, όπω στην περίπτωση αυτή, διότι δεν είναι πλέον πολιτικό πρόβλημα, διότι οι συνθήκε είναι ξεκάθαρε αν να τι αρμοδιότητε του ΔΕ. Αλλά θα πρέπει να πούμε πω τόσο το Συμβούλιο αλλά και η Κομισιόν χρειάζεται να αναλάβουν τι ε, δεσμεύσει του ε, μετά από την έγκριση της Λισαβόνας και να σεβαστούν τις ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και τις σχετικές εξουσίες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να είχαν πετύχει. Και το τονίζουμε αυτό το ζήτημα, επαναλαμβάνοντα λοιπόν όχι μόνο τις ευχαριστίες μου που ήρθατε δύο φορές, αυτή είναι η τρίτη στην ουσία που παρίσταται ενώπιον μας ε, και σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να συνεργαστούμε προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το είπατε και εσείς επανειλημμένα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε χέρι-χέρι για να μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε οι μεν τους δε ως εχθρούς, ως αντιπάλους, αλλά ως συνεργάτες. Γι' αυτό λοιπόν επιθυμώ αυτή τη θέση να έχετε και εσείς στο Συμβούλιο και εσείς προσωπικά Πρόεδρε και σας δίνω το λόγο για να μας μιλήσετε σχετικά με τις προτεραιότητες σας. Ευχαριστώ. Ačiū. Ε, Gerbiamas pirmininkė, gerbėmėjai parlamentai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Η Λιθουανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην Επιτροπή αυτή για να κάνω μια παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής. Να παρουσιάσω συγκεκριμένα το πρόγραμμα της Προεδρίας στον τομέα της Αλίας. Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα έχουμε 28 μέλη μετά την ένταξη της Κροατίας, είναι ιστορική πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα μου ευκαιρία να δείξουμε ότι μια μικρή χώρα μπορεί να λύνει προβλήματα αποτελεσματικά και με τρόπο ποιοτικό. Είναι αυτή μια ευθύνη που απολαμβάνουμε, για την οποία είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να είμαστε έντιμος διαμεσολαβητής στη λήψη των αποφάσεων και θα συμβάλλουμε ώστε να ε, υπάρχει συνέχεια στις διαδικασίες και να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εταίροι. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική προεδρία προσανατολισμένη προς την επίτευξη αποτελεσμάτων για να επιτύχουμε τους στόχους μας μιας αξιόπιστης και ανοιχτής αναπτυσσόμενης Ευρώπης. Μία πρόκληση για μένα ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου είναι να συνεργαστώ μαζί σας επικοδομητικά και παραγωγικά. Με εσάς που είστε συνομοθέτης και εταίρος ώστε να διασφαλίσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα από το έργο που επιτελούμε για τους πολίτες μας. Οι τελευταίοι απαιτούν να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο και να δουλέψουμε με προσανατολισμό τα αποτελέσματα σε θέματα σημαντικά όπως η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και άλλα πιο βραχυπρόθεσμα θέματα, ιδιαίτερα ε, σε εποχές οικονομικής κρίσης για τους πολίτες ε, αυτή τη δύσκολη περίοδο. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας, καθώς θα προχωρούμε την πολύ σημαντική νομοθετική μας ατζέντα, το θεματολόγιό μας και έχω δώσει οδηγίες στους συνεργάτες μου να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή αυτή. Καταρχήν, να αναφέρω τις γενικές προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας εστιάζει στη δημιουργία μιας Ευρώπης αξιόπιστης, αναπτυσσόμενης και ανοιχτής. Είναι ένα πρόγραμμα συνεκτικό που καλύπτει την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, την οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη, απασχόληση ιδιαίτερα των νέων, επίσης την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την περιφερειακή ε, ασφάλεια και το περιφερειακό άνοιγμα. Ο προεδρεύων στο Συμβούλιο Γεωργίας και Ελίας έχω ένα όραμα. Να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένας τομέας βιώσιμος στην αλληλεία, ο οποίος θα είναι και ανταγωνιστικός, σύγχρονος, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των αποθεμάτων και την προστασία τους. Πριν επισέλθω στις λεπτομέρειες του προγράμματος Προεδρίας στον τομέα της Αλίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου, τον κύριο Σάιμον Κόβενι, για το εξαιρετικό έργο του και για τη φιλοδοξία του να επιτύχει συμφωνία μαζί σας σχετικά με το βασικό κανονισμό και την κοινή οργάνωση της αγοράς. Πρόκειται για εξέχον επίτευγμα που δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση. Είναι ένα ε, ε, εξαιρετικό παράδειγμα πολιτικής ηγεσίας και υπ' αυτή την έννοια θέλω να ευχαριστήσω και τους συζηγητές... Ε, Ρόντους και Σίβενσον και των ε, Σκιωδών και θέλω να ευχαριστήσω και σας κύριε Πρόεδρε για την ε, συμβολή σας σε αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα. Είμαι βέβαιος ότι με την απαραίτητη πολιτική βούληση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το ίδιο επί... θετικό αποτέλεσμα και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλληλεία. Και τώρα θα στραφώ στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του Προεδρίας μας στον τομέα της Αλληλείας. Θέλω να διακρίνω δύο σειρές προτεραιοτήτων. Η πρώτη είναι να επιτευχθεί πρόοδος ε, σε σχέση με αυτό το Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλληλεία, το οποίο είναι στον τρίτο πυλώνα της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Η δεύτερη σειρά προτεραιοτήτων σχετίζεται με το γεγονός ότι τώρα είμαστε στο δεύτερο εξάμεινο και πρέπει να υιοθετήσουμε αποφάσεις για το 2014 για τα ΤΑΚ και τις προτάσεις για τις ποσοστώσεις, δηλαδή και τα ΤΑΚ, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Η προτεραιότητα οι μας ε, γιατί στη μεταρρύθμιση θα είναι να επιτύχουμε πρώτη, συμφω... Ε, πρώτη ανάγνωση συμφωνία μαζί σας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλία. Όπως γνωρίζετε, από πέρσι τον Οκτώβριο έχουμε καταρτήσει μια μερική γενική προσέγγιση από πλευράς Συμβουλίου. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια πλήρη γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Και όταν είναι έτοιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαπραγματευθεί, θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Τώρα, ποια είναι τα άλλα θέματα ε, που πρέπει να λυθούν στο Συμβούλιο είναι τα κονδύλια για το Ταμείο. Πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το ταχύτερο δυνατόν το Ταμείο αυτό και γι' αυτό επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει τις προτάσεις στην Ολομέλεια και να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Γνωρίζετε καλά ότι μεγάλο κομμάτι, για να μην πω ολόκληρο το δεύτερο εξάμεινο, το Συμβούλιο θα απασχοληθεί με την ευθύνη που έχει να προετοιμάσει και να αποφασίσει επί των διαφορετικών τάκ και ποσοστώσεων για τον επόμενο χρόνο. Τέσσερις αποφάσεις πρέπει να ληφθούν φέτος. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να φροντίσουμε του χρόνου να γίνει ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο επί της ε, ανακοίνωσης της Επιτροπής Διαβουλεύσεις για τις αλληλευτικές δυνατότητες το 2014. Η ανακοίνωση παρουσιάζει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά πολλά μένουν ακόμη να γίνουν στον τομέα αυτών. Καταρχήν πρέπει να αναφέρω ότι το 80% των αλλιευμάτων που καλύπτουν 41 διαφορετικά αποθέματα ξέρουμε ποια, ποιο είναι η μέγιστη ε, βιώσιμη απόδοση για αυτά για πάνω από το 60% αυτών των αποθεμάτων μπορούμε να πούμε ότι ήδη αλλιεύονται ε, δύο χρόνια μπροστά από το στόχο. Δηλαδή ο στόχος έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση δύο χρόνια πριν από αυτό που πρόβλεπε ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να εφαρμοστεί το σύστημα ε, MSY, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, το 2015, όπου αυτό θα είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσω να ε, στηριχθώ, να αξιοποιήσω αυτό το, αυτή την ενθαρρυντική τάση και θα στηριχτώ και στη σκληρή δουλειά των προκατόχων μου. Επίσης, ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία έχουμε ήδη ε, ποσοτικά προσδιορισμένη επιστημονική ε, ε, τεκμηρίωση έχει αυξηθεί πολύ και αυτό είναι σημαντικό γιατί μας δίνει δεδομένα για να λάβουμε αποφάσεις. Τρίτον, η αλλιευτική προσπάθεια έχει μειωθεί σημαντικά και αυτό μειώνει την αλλιευτική πίεση στα αποθέματα ηχθείων, πράγμα που με τη σειρά του τους επιτρέπει να ανανύψουν και να αυξηθούν. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα αποθέματα στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα είναι σε καλή κατάσταση, ενώ στη, στα δυτικά ύδατα και τα ύδατα της Ιβηρικής, όπως και τη Μεσόγειο και τη, τον Εύξηνο Πόντο, εκεί χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να βελτιωθούν τα αποθέματα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα ΤΑΚ πρέπει να λάβει υπόψη τρεις αρχές. Πρώτον, να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμα διαχειριστικά προγράμματα όπου υπάρχουν. Δεύτερον, να εφαρμοστεί άμεσα το σύστημα MSY της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ε, όπου αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε το ΤΑΚ, τα ΤΑΚ και τρίτον, θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε κοινωνικο-οικονομικά θέματα, διότι οι αλληλείς πρέπει να ε, μπορούν να έχουν ένα βιοποριστικό επάγγελμα, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Η... Σε σχέση με τα τάκ, το Συμβούλιο πρόκειται να κάνει τα εξής. Θα καταπιαστεί με την Αντσούγια τον Ιούλιο, τα τάκ της Βαλτικής τον Οκτώβριο, τα τάκ, τα ε, μέγιστα επιτρεπόμενα λεύματα για τον εύξηνο πόντο το Δεκέμβρη και τα βασικά ΠΑΚ το Δεκέμβριο. Τώρα, ε, για τις άλλες προτάσεις. Καταρχήν η απαγόρευση της ε, απόρριψης στη θάλασσα, ο κανονισμός Omnibus, σαν πολυκανονισμός. Μια άλλη προτεραιότητα στη συνόδους του Συμβουλίου είναι η συζήτηση επί των κανονισμών αυτών και προσβλέπουμε στην εφαρμογή της απαγόρευσης της επαναπόρριψης. Περιμένουμε και τις προτάσεις της Κομισιόν για τις απαραίτητες τροπολογίες στην υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία είναι πολύ σημαντική, οπότε θέλουμε να αρχίσουμε να εργαζόμεθα επ' αυτή στο ταχύτερο δυνατόν. Οι Υπουργοί θα επιδιώξουν μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης ήδη στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την ευθυγράμμιση της κειμένης νομοθεσίας προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας ε, την πρόταση για την ευθυγράμμιση των τεχνικών μέτρων στην Μεσόγειο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμπεριλάβουμε και άλλες προτάσεις, ε, ίσως για τα κοιτοειδή αλλά ο χρόνος πιέζει και πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας και να ομολογήσω ότι δεν είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Λιθουανική Προεδρία θα εργαστεί μαζί σας ε, κατά την Προεδρία της για να έχουμε ένα γνήσιο διάλογο επί των μακροπρόθεσμων διαχειριστικών σχεδίων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε διαφωνίες και τριβές μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ε, τα προηγούμενα τρία χρόνια. Καταλαβαίνω απόλυτα τη σοβαρότητα αυτού του θέματος για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα διαχειριστικά σχέδια αποτελούν μια επιτυχία στην κοινή ελληνική μας πολιτική. Όπου είναι σε ισχύ ε, διαχρονικά βελτιώθηκαν τα αποθέματα και ως εκπρόσωπος μιας βαλτικής χώρας μπορώ να αναφέρω το παράδειγμα του ε, ε, βακαλάου στην Ανατολική Βαλτική. Γι' αυτό τα μακροπρόθεσμα διαχειριστικά προγράμματα, σχέδια είναι κρίσιμα ε, ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμης αλίας στα ενωσιακά ύδατα. Ε, ξέρουμε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει και πολύ καλή θέληση για να βρεθεί μια κατάλληλη λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Και πράγματι υπάρχουν δύσκολες πλευρές σε αυτό το θέμα που δεν επιλύονται εύκολα. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ε, υπόθεση και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα αποθέματα Βακαλάου. Ε, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Στις αρχές του χρόνου οι υπουργοί σχεδόν ομόφωνα ανακοίνωσαν ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης θα παραμείνουν στοιχεία κλειδί στη βιώσιμη διαχείριση ε, της αλληλίας και ενώ συζητούσαμε για τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ανέλαβε την υποχρέωση το Συμβούλιο να συνεργαστεί με Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέβρεση μιας λύσης η οποία θα σέβεται τις νομικές θέσεις και των δύο πλευρών, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η κατάρτιση πολιετών σχεδίων κατά τη νέα περίοδο μετά την μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ε, υπάρχει και μια διοργανική ειδική ομάδα, task force, η οποία μπορεί να ε, αναλάβει να εξετάσει περισσότερο το θέμα αυτό. Το φθινόπωρο είναι πολύ, πολύ άσχολη εποχή για την εξωτερική πολιτική αλληλεία. Στο Συμβούλιο θα έχει ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο για την προετοιμασία των ετήσιων διαβουλεύσεων με την Ορβηγία και τις προετοιμασίες για την ε, ετήσια σύνοδο ICAT. Τώρα, εις ό,τι αφορά τις εταιρικές συμφωνίες για την Ελία, τα βασικά θέματα είναι η Μαυριτανία και το Μαρόκο. Τώρα, ε, για την Μαυρετανία. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου αν θα εγκρίνει δηλαδή ή όχι ένα νέο πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με τη Μαυρετανία. Αν το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει με το πρωτόκολλο αυτό, θα υπάρξουν ενδεχομένως πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους στόλους σε εκείνα τα ύδατα και θα υπονομευθούν και οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρωτόκολλο στο μέλλον. Η Λιθουανική Προεδρία αναγνωρίζει ότι οι αλλιευτικές δυνατότητες έχουν μειωθεί και τώρα οι τεχνικές προϋποθέσεις και όροι για το νέο πρωτόκολλο είναι πιο αυστηροί και μπορεί να είναι απογοητευτικοί από οικονομική άποψη όμως είναι εποφελής ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διατήρηση των αποθεμάτων. Κάποιες βελτιώσεις έχουν ε, υπάρξει ε, από την Κοινή Επιτροπή το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο που έγινε η τεχνική συνάντηση. Τώρα, για το Μαρόκο, ο αλλιευτικός στόλος ε, περιμένει ανυπόμονα τις αποφάσεις που θα απαλείψουν τα εμπόδια για την υπογραφή του νέου πρωτοκόλλου και ο τομέας ζητεί την επίτευξη συμφωνίας το ταχύτερο δυνατόν. Και εδώ παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών προτεραιοτήτων στον τομέα της Αλίας επί Λιθουανικής Προεδρίας. Είναι καινούρια πρόκληση για μας κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα όταν το θεματολόγιο μας περιλαμβάνει τόσα πολλά θέματα και όταν οι προσδοκίες είναι τόσο μεγάλες για μια πραγματική αλλαγή στην κοινή ελληνική πολιτική. Φέτος είναι το έτος των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να θυμόμαστε ότι συμμεριζόμεθα μια κοινή ευθύνη υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να ε, συνεργαστούμε χέρι-χέρι προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, τώρα Είμαστε στο επίκεντρο της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ελπίζω να συνεργαστούμε μαζί αποτελεσματικά, επικοδομητικά. Ελπίζω ότι μας ενώνει ένας κοινός στόχος, δηλαδή να ολοκληρώσουμε τις ε, βασικές μας εργασίες και να πραγματοποιήσουμε αυτά που πρέπει πριν από το 2014 και πριν από τις εκλογές του, για το Κοινοβούλιο του χρόνου για να εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον στις θάλασσές μας και τους αλληλείς μας. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ευτυχής να δεχτώ τις ερωτήσεις από εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Φυσικά πολλές ερωτήσεις. Θα κάνουμε έναν γύρο παρεμβάσεων θα αρχίσουμε με τους συντονιστές και μετά οι υπόλοιποι βουλευτές, επειδή οι συντονιστές είχαν ήδη τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ μας, μεταξύ σας θα λάβουν το λόγο αργότερα και οι βουλευτές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό που ήρθε και πριν ζήτησα το λόγο. Τώρα όμως σας άκουσα πολύ προσεκτικά γιατί παρουσιάσατε όλο το πρόγραμμα εργασίας σας και καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βασική σας πεποίθηση υπέρ των μακροπρόθεσμων διαχειριστικών σχεδίων γιατί τόσο ξεκάθαρη γλώσσα δεν έχω ακούσει από κανένα υπουργό του Συμβουλίου πόσο σημαντικά είναι σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Υπενθυμίζω όμως αυτά τα πλαίσια ότι στους τριμερείς διαλόγους για το βασικό κανονισμό σε αυτό το θέμα συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να συστήσουμε ένα task force, μια ειδική ομάδα με συμμετοχή και των τριών θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι ε, είναι καθήκον δικό σας ε, επίση να το υποστηρίξετε αυτό και μάλιστα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι θα το κάνετε γιατί και εσείς είστε πεπισμένος ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση και για τους αλληλείς και για τα ψάρια. Να έχουμε δηλαδή μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Θέλω επίσης να σας καλέσω να ασχοληθείτε με την αλληλεία ε, ανοιχτής θαλάσσης γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου. Κατά τα άλλα, σας ε, είπα και πριν τα θέματα που με απασχολούν και δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο από τους συναδέλφους μου. Η κυρία Λοβέν, ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και πάλι τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα ήθελα να θέσω σε σχέση με τις προτεραιότητες σας. Πρώτον, δεν ανέφερα προηγουμένως ότι ήμουν εισηγήτρια της εξωτερικής διάστασης, οπότε επικριτώ το γεγονός ότι έχετε ως προτεραιότητά σας να εξασφαλίσετε ότι οι συμφωνίες με το, με το Μαρόκο και την Μαυριτανία ε, θα προχωρήσουν ε, όπως πρέπει και να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο συγγνώμη, ε, υπήρξε πολύ σαφές σε σχέση με αυτά που ήθελε ε, για το μέλλον αυτών των ε, αλληλευτικών συμφωνιών ε, των βιώσιμων. Μάλιστα υπάρχει και ένας νέος τίτλος ε, για ε, αυτές τις συμφωνίες στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει πλεόνασμα αλλιευμάτων που δεν τα χρειάζεται ο τοπικός πληθυσμό και άλλο ένα στοιχείο είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία το Κοινοβούλιο έχει τονίσει πολλές φορές και εάν δεν γίνονται σεβαστές αυτές οι πολύ σημαντικές αρχές, το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του σε καμία από αυτές τις αλληλευτικές συμφωνίες στο μέλλον. Επίσης, θα ήθελα δύο ερωτήματα να σας θέσω, διευκρινήσεις μάλλον, σε σχέση με αυτά που είπατε. Αν πρόκειται θα να ασχοληθείτε με ε, το θέμα της ανοιχτής, ε, της, θάλασσας, ε, της ανοιχτών θαλασσών, το είπε και η κυρία Ρόνταστ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το θέμα. Έχει υποβληθεί πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολύ καιρό και εξ όσων γνωρίζω το Συμβούλιο δεν το έχει καν συζητήσει στην πρώτη φάση καν. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πότε θα γίνει αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στο Omnibus, Αναφερθήκατε στις απορρίψεις, ε, στην απαγόρευση απορρίψεων και την εφαρμογή. Ε, αλλά δεν μιλήσατε για, για τις δοκιμές ε, που πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν ήδη από την επόμενη χρονιά και θα ήθελα να μας πείτε πώς ε, θα, πώς θα προχωρήσει αυτό. Για τα συνολικά επιτροπόμενα λιεύματα και τις ποσοστώσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έτος γιατί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίσει ε, τα ποσά αυτά για να επιτύχει τους στόχους ε, ώστε να επιτρέψει στα ε, αλλιευτικά αποθέματα να φτάσουν σε επίπεδα πάνω από αυτά ε, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης μέχρι το 2015. Οπότε θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην, ε, στον, για τον καθορισμό φιλόδοξων ποσοστώσεων αυτή τη φορά. Κατά πάσα πιθανότητα ε, θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο που έχουν συμφωνήσει ε, τα δύο όργανα. Ελπίζω ότι θα το πετύχουμε και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να παραμείνετε κατηγορηματικός γιατί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε μέχρι το 2015 πρέπει να είναι φιλόδοξες οι ποσοστώσεις και θα ήθελα να υπενθυμίσω και και στην Προεδρία αυτό που αποφασίσαμε εμείς ε, μεταξύ μας ε, ότι δεν είναι δυνατόν ε, να πετύχουμε τίποτε αν ζητήσετε κάτι λιγότερο φιλόδοξο από αυτό που είχαμε συζητήσει. Όσον αφορά τώρα τα μακροχρόνια σχέδια διαχείρισης, θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα και για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σάντζε Περσέδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω με τη σειρά μου τον ε, Πρόεδρο του Συμβουλίου και να του ευχηθώ καλή επιτυχία και να τον ευχαριστήσω για την συνεργασία που δήλωσε πως θα έχει μαζί μας ε, σε θέματα μεταρρύθμισης στον Αλία και να αναφερθώ στην εξωτερική διάσταση και να θίξω το ζήτημα της Μαυριτανίας. Το Κοινοβούλιο πάντως δεν έχει εγκρίνει το ψήφισμα και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μια μετάθεση της απόφασης, αλλά με τη βούληση προκειμένου να δηλώσουμε στις μαυριτανικές αρχές πως ε, υπάρχει μια κάποια ανισορροπία στο ισχύον πρωτόκολλο, πρωτόκολλο και θεμητές ανησυχίες από πλευρά των ε, εκπροσώπων στην Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να επιληθεί. Θα πρέπει, χρειάζεται λοιπόν να αποφεληθούμε του χρόνου προκειμένου να επιληθούν τα εκρεμή ζητήματα διότι στόχος ε, είναι φυσικά να συνεχίσει η αλία στην περιοχή και να μην ε, μειωθούν οι δυνατότητες αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της ε, Επιτροπής Αλίας του Ευρωκοινοβουλίου και να συμβάλλει στην επίλυση του όλου προβλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάντσο Πιστεύω. Κύριο Στίβενσον έχει το λόγο. Αντιπρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ε, να καλωσορίσω γενικώ τη Λιθουανική Προεδρία. Σας συναντήσαμε για γεύμα στην ε, πρεσβεία ε, πριν από μερικέ ημέρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρετε το θέμα των πολιετών προγραμμάτων. Βέβαια, είστε η 8η Προεδρία που το κάνει αυτό. Οι προηγούμενε 7 Προεδρίε χαρακτηρίστηκαν από αυτέ που υποσχέθηκαν πολλά και δεν πέτυχαν τίποτα και κάποιες άλλες που πάλι δεν πέτυχαν τίποτα. Ε, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω τι το ιδιαίτερο έχετε σκοπό να κάνετε. Κάτι ακόμη. Συμφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εξακολουθεί να υπάρχει υπεραλίευση του ενωσιακού στόλου και αν συμφωνείτε πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε ε, τα χρήματα των φορολογούμενων για ε, την κατασκευή νέων αλλιευτικών σκαφών. Ευχαριστώ. Gracias, señor Señora García κυρία Γέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ και να σας παροτρύνω προκειμένου να συνεργαστείτε στενά μαζί μας και να γνωρίζετε ότι θα τύχετε τη στήριξη των Ισπανών Σοσιαλιστών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου του σας. Συμφωνώ μαζί σας, μια μικρή χώρα μπορεί να συμπεριλαμβάνει άτομα ιδιαίτερα ικανά και να είναι σε θέση να πετύχουν πολύ περισσότερα από ότι μια χώρα πολύ μεγαλύτερη. Δεν πρόκειται για εδάφη, πρόκειται για πρόσωπα, για άτομα. Και εσείς ε, αναφέρατε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να επιτευχθεί με πάση προσπάθεια όπως συνέβη και με την προηγούμενη Προεδρία που ήταν ε, ιδιαίτερα αποτελεσματική και ε, προώθησε ε, μια σειρά τριμερών διαλόγων. Επίσης να σας κάνω και ένα αίτημα Δεν χρειάζεται να σας πω εσείς πρέπει να δεσμευτείτε περισσότερο, αλλά να ε, εννοείτε αυτά που λέτε για να τα μεταφέρετε σε πράξη. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα είναι αυτή, στην ε, Ευρώπη είναι το θέμα της οικονομικής ύφεση, κάτι το οποίο δημιουργεί περισσότερη φτώχεια, λιγότερες ε, θέσεις εργασίας, ε, περισσότερη ανεργία και λιγότερες ευκαιρίες ε, στον τομέα της αλίας. Η χώρα μου είναι μια χώρα που ασχολείται ιδιαίτερα με την ε, αεραστεχνική αλία και αυτό είναι αυτό το οποίο μας ανισχύει ιδιαίτερα διότι αυτό επηρεάζει τον χαρακτήρα της ε, αλίας. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε το σχέδιο ενός ψηφίσματος για ένα ταμείο και ο ρόλος ε, που θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαδραματίσει προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους νέους να μπορέσουν να ενταχθούν στον κλάδο και να υπάρξει μια συνέχιση αυτής της αλίας που όχι μόνο προϋποθέτει κάτι και μάλλον ε, αποτελεί μια προσφορά στο ΑΕΠ των μεσογειακών χωρών αλλά προϋποθέτει και μια κουλτούρα ε, προϋποθέτει κάποια ήθη και έθιμα που όλες όλοι οι Ευρωπαίοι του Βορρά και του Κεντρικής Ευρώπης θέλουν κάποια στιγμή να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη επίσης ότι οι Ισπανοί είμαστε οι πρώτοι καταναλωτές και μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός πως όταν μιλούμε για εξωτερική πολιτική και την αγορά προϊόντων αλίας από τρίτες χώρες πρέπει να τους ζητάμε τις ίδιες προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που απαιτούμε από τους δικούς μας. Λοιπόν, η σήμανση και οι ετικέτες που, που επιτίθενται σε αυτά τα προϊόντα τα αλληλευτικά είναι ελλειπή σε σχέση με αυτές που επιβάλλουμε στους δικούς μας ελεύθερους. Τώρα, σε ό,τι φορά το Μαρόκο, είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι για πάνω από 1,5 χρόνο μικροί αλληλείς οι οποίοι δεν έχουν άλλο μέσο επιβίωσης ε, είναι το μόνο τους βιοπαριστικό έργο δεν εφαρμόζουμε λοιπόν τους ε, ίδιους κανόνες που, έχουμε, που εφαρμόζουμε μάλλον ακόμα και στις αγορές μας από την Ταϊλάνδη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε το ζήτημα των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα τη Αλίας. Ευχαριστώ και τον για το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, βόντα να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας και προφανώς όλα τα μέλη θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας για να δοθεί καλή συνέχεια στο αξιέπαινο πρόγραμμα σας. Τώρα τα μακροπρόθεσμα διαχειριστικά προγράμματα και παραθέτω εσάς είναι εργαλείο για τη βιωσιμότητα. Α, όντως έτσι είναι. Είναι σημαντικά όπως ο βασικός κανονισμός αφού είναι εργαλείο για τη βιωσιμότητα. Πάντως νομίζω ότι ε, ε, θέλετε να κάνετε το σωστό και είναι κρίμα που στα πέντε χρόνια της εντολής μας εμείς δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε τίποτε εδώ. Ε, αυτό μας δημιουργεί μια αμηχανία. Ελπίζω να συνεργαστούμε και ελπίζω και η ειδική μονάδα αυτή, η ομάδα της Task Force να ασχοληθεί. Ελπίζω να παρακολουθήσετε από πολύ κοντά την κατάσταση σε σχέση με την ε, μη βιώσιμη αλληλεία και τις κυρώσεις, γιατί δεν μπορεί η Κομισιόν να κατηγορεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ότι δεν είναι στο πλευρό της, γιατί ο προκατοχός σας σε παρουσία της Επιτρόπου μας είπε ότι είναι μαζί μας το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει νομίζω Συμβούλιο που θα είναι κατά της εφαρμογής εμπορικών κυρώσεων όταν υπάρχει ε, άναρχη Και ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε την κατάσταση εκεί και ελπίζω αργότερα να ακούσουμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα από την Επίτροπο. Επίσης θέλω να σας επενέσω για μία αναφορά που κάνατε στην αρχική σας ε, παρέμβαση όπου αναφέρατε τη σημασία των κοινωνικο-οικονομικών θεμάτων γιατί η αλληλεία γίνεται κυρίως σε περιοχές χωρίς εναλλακτική απασχόληση και πάντα πρέπει να βρούμε ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας ε, και οικονομικών και κοινωνικών ε, και κοινωνικών παραγόντων και χαίρομαι πολύ και σας συγχαίρω που το αναφέρατε. Ε, άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριε Πρόεδρε έχει το λόγο μια που κάποιος άλλος δεν υπάρχει προς τον παρόν που θέλει να το λόγο. Ε, ε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας, για όλες τις ερωτήσεις που θέσατε. Σημείωσα τα πάντα και θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη ε, κατά τους ερχόμενους έξι μήνες. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για τις ευχές σας, ε, για την Προεδρία μας και θα προσπαθήσω τώρα σύντομα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Η κυρία Λουρίκε Ρόνταστ με ρώτησε για τα ε, μακροπρόθεσμα ε, διαχειριστικά προγράμματα και μας μιλήσατε επίσης και για την Task Force, την ειδική ομάδα δράσης. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας για αυτό το θέμα, για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα και θα υποστηρίξω αυτή την πρωτοβουλία στο Συμβούλιο. Μαζί με την ομάδα μου θα, προσπαθούμε να βρούμε, προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες ε, λύσεις. Τα πολιετή προγράμματα βέβαια είναι ένας από τους κύριους στόχους της ε, μεταρρύθμισης. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό να επιληθούν τα εκκρεμή ζητήματα. Πρέπει να ε, περάσουμε την έγκριση των προγραμμάτων. Καλή θέληση να υπάρχει και νομίζω θα τα καταφέρουμε μέσω των συζητήσεων. Πολλές προηγούμενες ε, προεδρίες προσπάθησαν, ε, κύριε Στίβενσον, να λύσουν τα θέματα αυτά. Ε, το είπατε κι εσείς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια ευνοϊκή θέση σε σχέση με την επίλυση του θέματος αυτού, γιατί έχουμε το βασικό κανονισμό τώρα για την μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Μιλούμε για την ε, διοργανική task force ε, που μπορεί να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό. Εγώ θα ήθελα τα ε, μέλη του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να επιτύχουμε τους συγκεκριμένους στόχους που έχουμε θέσει. Τώρα, όσον αφορά την αλληλεία ανοιχτών θαλασσών και την επίβλεψη στον τομέα αυτών. Εμείς ε, ακούσαμε τα αποτελέσματα από τους αμπειρογνώμονες και από τη δημόσια ακρόαση που οργανώθηκε. Συμφωνώ. Το Συμβούλιο συνομοθέτης πρέπει να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη συζήτηση του θέματος αυτού. Να ευχαριστήσω ε, τον ε, κύριο Αρσένη και την κυρία Ρόντας ε, για την επιστολή τους, στην οποία εξέφρασαν την ανησυχία τους για το θέμα αυτό. Η Λιθουανική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και θα προγραμματίσουμε τα πράγματα εγκαίρως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική διάσταση της ε, αλλιευτικής πολιτικής, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της εξωτερικής ε, διάστασης και την ε, αναγκαιότητα των διατάξεων και των όρων στους οποίους αναφερθήκατε. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στο βασικό κανονισμό της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής και θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τις αρχές αυτές. Όσον αφορά τώρα το στενό του Σκάγκαρακ, κυρία Λέβιν, Ελπίζαμε να, υπήρξε, να, υπάρχει κάποια, να, να υπήρχε κάποια λύση κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Τώρα βέβαια θα προσπαθήσουμε εμείς να επιμείνουμε, να εντείνουμε στις προσπάθειές μας ε, για να αρχίσουμε ε, συναντήσεις τριμερούς ε, διαλόγου το φθινόπωρο και να καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία και σε αυτό. η αηφορία είναι βεβαίως ε, βασικός ε, στόχος και με την ε, πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση και την έγκαιρη εφαρμογή της, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε βιώσιμη αλία στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτό, είναι, αυτό προσπαθούμε όλοι να πετύχουμε για τη συμφωνία μας τώρα με την Μαυριτανία. Ε, Καταλαβαίνουμε ότι το πρωτόκολλο τώρα και οι αλευτικές ε, δυνατότητες που έχουν συμπεριληφθεί δεν είναι ελκυστικά, δεν, δεν είναι οικονομικώς τόσο ελκυστικές όσο θα μπορούσαν να είναι. Είναι πολύ πιο αυστηρές, όμως χρειάζονται όσον αφορά την διατήρηση των ηχθιαποθεμάτων. Η τροποποίηση του πρωτοκόλλου μας δίνουν ε, την ελπίδα ότι θα είναι για τους Ευρωπαίους αλληλείς πιο ελκυστική η αλληλεία ε, στην περιοχή Πρέπει όμως να μην μας διαφεύγει ότι ειδικότερα ως προς τα ε, βενθοπελαγικά είδη ο αλλιευτικός μας ε, στόλος δεν έχει άλλες δυνατότητες ε, στα, στα δυτικά της Αφρικής. Και σε σχέση τώρα με το ερώτημα ε, για το ταμείο του κυρίου Στίβενσον θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο μετά από μεγάλες συζητήσεις ε, ενέκρινε την απόφαση του τον Οκτώβριο του 2012 και η κατασκευή νέων αλληλευτικών σκαφών ε, δεν ε, συμπεριλήφθηκε στις υποψήφιες δράσεις. Όταν θα είναι σαφή η θέση, η θέση και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα προβούμε στι διαπραγματεύσει για να δούμε ποιε είναι οι αποδεκτές θέσει ε, των δύο συνομοθετών ε, για ε, τις επιλέξιμες δράσεις, τις επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο αυτό. Όσον αφορά την παράκτη αλία, πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας. Είναι γεγονός ότι η αλία μικρής κλίμακας, η ερασιτεχνική αλία, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντικό εισόδημα για τις παράκτιες κοινότητες και συνήθως είναι βιώσιμη αυτή η αλία. Οπότε πρέπει να την υποστηρίξουμε και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξεύρουμε ε, κονδύλια στο Ταμείο Αλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων. Η αλληλεία αυτή ε, διαφέρει βέβαια ανάλογα με το σημείο ε, της Ευρώπης ε, για το οποίο μιλούμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ότι πρόοδος θα σημειωθεί σε όλα τα προβλήματα αν συνεχίσουμε τη συνεργασία και αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αναζητήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ολοκληρώνοντας, μερικές ακόμη σκέψεις όσον αφορά τη μακροαλία. Το Συμβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση εδώ και κάποια χρόνια και είμαστε απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να βρούμε μία λύση. Και υπάρχει περαλίευση του σκουμπριού. Νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν εμπορικές κυρώσεις ε, εναντί των χωρών που υπεραλλιεύουν. Αλλά το Συμβούλιο δεν είναι απολύτως υπεύθυνο, είναι στα χέρια της Επιτροπής ε, το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας πει ε, τα, ε, τις τελευταίες εξελίξεις ε, στον τομέα αυτό. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα μία ακόμη φορά να πω ότι πάντοτε θα αξιολογούμε το σημαντικό ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην νομοθετική διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε να ε, συμμετέχουμε σε επικοδομητικό διάλογο ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσω συζητήσεων ε, και συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι, κάποιο σχόλιο. Όχι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για μια ακόμα φορά και ελπίζουμε αυτές οι αμοιβές υποσχέσεις περί συνεργασίας να υποδοθούν. Ευχαριστώ. Είστε ελεύθερος. cuestión antes de que, según el orden del día, Σύμφωνα με τη διάταξη, σήμερα το πρωί εγώ έκανα κάποιο λάθο και δεν εγκρίναμε τα πρακτικά τη συνεδρια ω έως 29-30 Μαΐου που ήταν στο σημείο 3 τη μεσέ διατάξεω. Είχαμε την ψηφοφορία, εγώ τα είχα λίγο χαμένα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εγκρίνουμε λοιπόν αυτά τα πρακτικά. Το επόμενο σημείο είναι ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Μαρία Δαμανάκη. Η συνεδρίαση αυτή πρόκειται να είναι ανοιχτή. Τελικά αποφασίσαμε να γίνει κερδισμένο των θυρών και ε, έπρεπε να ξεκινήσει στις 4 και 30, 16 και 30. Ως εκ τούτου έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας ε, πάνω κάτω. Θέλετε να πάρετε να πιείτε ένα καφεδάκι να ξεμουδιάσετε εκτός, εκτός, αλλά ο Ριμπελίνη δεν είναι εδώ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλο σημείο της μέσης διατάξεως. Το ζήτημα είναι ότι... Αλλά ο Σάντσος Πεσέδο είναι εδώ, έτσι δεν είναι. Αν θέλετε θα μπορούσαμε να περάσουμε στο ζήτημά σας κύριε Σάντσος Πεζέδο στο σημείο 11 για να ξεμπερδεύουμε και να τελειώσουμε και έτσι νωρίτερα το απόγευμα. Ο εισηγητή είναι εδώ, δεν ξέρω αν στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψε, να δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν έχω πρόβλημα σε ό,τι με αφορά να εξετάσουμε τώρα το ζήτημα. Συγγνώμη, συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος συμφωνεί η Επιτροπή να περάσουμε στην εξέταση του σημείου 11. Η Κομισιόν είναι παρούσα? Όχι. Δεν είναι παρούσα η Κομισιόν. Δεν έχουμε κανέναν από την Κομισιόν, άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων ε, που αφορά στις τροπολογίες, έτσι δεν είναι. σχετίζεται με τις τροπολογίες πάντως. Είναι η ανταλλαγή με την Κομισιόν. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να παρίσταται η Κομισιόν, εντάξει. Τώρα για τις τροπολογίες και σαν τους Πρεσέδο, παρακαλώ, πείτε τα μας όλα. Ναι, πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών. Είδα πως εδώ οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ε, έχουν κατευθεί από πλευρά ε, συναδέλφων εκτό από τον κύριο Αλκαντέκ, ο οποίο δεν βρίσκεται εδώ. Να ζητήσω τον κύριο Τόμα, τον κύριο Πατράου Νέβε ε, και τον ε, κύριο Κάλαχερ. Θα του ακούσω λοιπόν και μετά να σχολιάσω επόμενα τι παρατηρήσει του και τα σχόλιά του. Gracias, señor Santipresidente. Ευχαριστώ κύριε Σάντσο Πεσέδο, κυρία Τόμα. Έχει το λόγο. Ε, es Υπάρχουν δύο ζητήματα. Εάν ε, λείπουν κάποιοι βουλευτές, ε, τι θα η υποχρέωση των βουλευτών είναι να είναι παρόντες, όχι να βρίσκονται εκτός αιθούση. Αυτό δεν με ανησυχεί. Αυτό που με ανησυχεί είναι περισσότερο το ζήτημα της Κομισιόν που δεν είναι παρούσα. Αλλά επειδή η συζήτηση αφορά στι τροπολογίε δεν είναι θεμελιώδη η παρουσία της Κομισιόν. Συνεχίζουμε λοιπόν την εξέταση του σημείου. Υπάρχουν ισχυρότερε ηγητέ. Κοιτάξτε, συνεχίζουμε τη συζήτηση ή όχι. Μένα το ίδιο μου κάνει. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Αλλά πείτε μου κάτι μην μένετε σιωπηροί ως ψάρια. δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει με τους ε, καταθέτες των τροπολογιών, διότι εγώ όταν έλαβα τα κείμενα δεν έλαβα και τις τροπολογίες ε, συγχρόνως και νομίζω ότι και οι συντάκτες των τροπολογιών δεν διαθέτουν τις ε, τροπολογίες. Δεν έχουμε λοιπόν, λοιπόν παρά να μεταθέσουμε την εξέταση του ζητήματο. Ναι. Κοίταξε δεν έχουν τώρα τροπολογίε, δεν τι έχουν σε μισή ώρα. Α, τι νομίζετε ότι θα είναι στη διάθεσή του, θα βρίσκονται στο γραφείο. Α, εντάξει, τότε α μην περιπλέκουμε τα πράγματα, μην δυσκολεύουμε τη ζωή μας, σταματάμε για 20 λεπτά. 4 25 θα είμαστε εδώ πάλι. Χαίρομαι που είμαι εδώ και πάλι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Να πω δύο λόγια πρώτα απ' όλα για τις προθεσμίες για, την υδατοκαλλιέργεια όπως μου ζητήσατε. Νομίζω ότι είναι αυτό από τα θέματα που η Επιτροπή ενδια... σας ενδιαφέρεται πολύ και διευκρινίζω ότι ο τομέας υδατοκαλλιέργειας είναι ένας τομέας που πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί από εμάς. Η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια θα μας βοηθήσει με, να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ζήτηση για τα θαλασσινά. Ο κλάδος υδατοκαλλιέργειας θα δώσει φρέσκα θαλασσινά υψηλής ποιότητα τοπικής παραγωγής ε, που θα συνάδουν με υψηλής ποιότητας πρότυπα θα δώσει και ανάπτυξη και απασχόληση και στις παράκτιες κοινότητες και στην ενδοχώρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να σπάσουμε τα εμπόδια και τους φραγμούς ε, που δεν επέτρεψαν να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια της Ένωσης και να δώσουμε στην πολιτική αυτή την ε, προσοχή που χρειάζεται. Προτεραιότητα, μείωση της γραφειοκρατίας, ε, απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς όμως να κάνουμε ε, πίσω και εκπτώσεις σε θέματα ζωτικά δεν θα πρέπει να συμβιβαστούμε σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα. Είμαι πεπισμένη ότι η υψηλή ποιότητα και η βιωσιμότητα πρέπει να είναι το ανταγωνιστικό μας βασικό πλεονέκτημα. Και έχουμε κάποια παραδείγματα στα κράτη-μέλη μας και τώρα είδα το καλλιέργεια, δηλαδή που μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο και την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Οι στρατηγικέ ε, προθεσμίες ε, για την υδατοκαλλιέργεια του Απριλίου ορίζουν το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόθεση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και αυτό που είναι τώρα υποχρέωση κάθε κράτους μέλους και αυτό είναι το καινοτόμο μέσο, τώρα ε, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ετοιμάσει εθνικό σχέδιο, ζητούμε από τα κράτη-μέλη δηλαδή να προετοιμάσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια που θα αντικατοπτρίζουν τις ε, ιδιαίτερες προκλήσεις και τα θετικά του στοιχεία. Η Κομισιόν θα βοηθήσει βέβαια να συντονίσει τις εθνικές δραστηριότητες και να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας και τα κράτη-μέλη όμως θα ετοιμάσουν τα εθνικά του σχέδια και η χρηματοδότηση θα στηρίζεται πάνω σε αυτά τα εθνικά σχέδια. Πρέπει να υπάρχει σαφές εθνικό σχέδιο. Αυτό θα είναι μια προϋπόθεση για να γίνει ε, συνέχιση της χρηματοδότησης. Θα υπάρχει ένα κονδύλιο για τη χρηματοδότηση, μια γραμμή στον προϋπολογισμό, ε, χωριστά για την υδατοκαλλιέργεια και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει ε, από αυτό το ταμείο. Τέλος, να σας ενημερώσω για, τη... για την οδηγική Ρέγκα και το σκουμπρί. Για τη Ρέγκα καταρχήν πρέπει να σας θυμίσω ότι οι Φερόες ε, βγήκαν από τη συμφωνία και μονόπλευρα αύξησαν την ποσόστοσή τους. Αυτή είναι μια απόφαση που την έλαβαν μονόπλευρα, εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποφάσισαν να αυξήσουν το μερίδιο των αποθεμάτων κατά 145%. 145%. Ενώ τα άλλα παράκτια κράτη, όλα και η Ρωσία και η Ισλανδία περιέκοψαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, περιέκοψαν κατά 23% τα μερίδια τους ως αποτέλεσμα της κακής κατάστασης του αποθέματος. Αυτά ε, είναι τα στοιχεία για να τα θυμάστε. Πρέπει να πείσουμε τις Φερόες ότι η απόφαση τους ήταν απαράδεκτη. Γι' αυτό το Μάιο η Κομισιόν άτυπα ενημέρωσε τις αρχές ότι η χώρα αναφέρονταν ε, ως χώρα που επιτρέπει την άναρχη αλληλεία και αν δεν διόρθωνε την κατάσταση μέσα σε ένα μήνα θα ίσχυαν μέτρα. Ένα μήνα αργότερα η, απόφα... η, απάντηση ε, από τις Φερόες έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αλλάξουν την απόφαση στην οποία εμένουν. Ίσως είδατε την αλληλογραφία αυτή. Μετά από διεξοδική ανάλυση, οι υπηρεσίες μου δεν πίστηκαν από τα επιχειρήματα που πρόβαλαν οι Φερόε, νήσι, και δεν είχαμε εναλλακτική από το να ε, θέσουμε σε εφαρμογή εμπορικές κυρώσεις. Να σας ενημερώσω εντωμεταξύ ότι οι ε, δανείοι υπουργοί, αλληλείας ε, εξωτερικών ήρθαν να με δουν. Και προσφέρθηκαν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ φερών και κομισιών. Ε, δέχτηκα με γνωμοσύνη προφανώς, γιατί πάντοτε πίστευα ότι το εμπορικό μέσο είναι η ίστατη καταφυγή και το πιστεύω αυτό, όταν όλα τα άλλα διαπραγματευτικά όπλα έχουν αποτύχει. Όμως από τότε δεν υπήρξε θετική αντίδραση από τις Φερόες νήσους, παρά τις προσπάθειες των δανεικών αρχών. Προσπάθησαν μεν, δεν υπήρχε αποτέλεσμα δε. Δεν είχα λοιπόν εγώ άλλη εναλλακτική από το να δώσω οδηγίες στις υπηρεσίες μου να προχωρήσουν και να επιταχύνουν την διαδικασία έγκρισης εμπορικών μέτρων. Και θα οριστικοποιηθεί νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα από τώρα αυτή η διαδικασία. Πάμε λοιπόν για τελική απόφαση τότε και θα εφαρμόσουμε το εμπορικό μέσο ε, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάω στο ε, Σκουμπρί που είναι το άλλο απόθεμα. Είχα ανταλλαγή ε, με τον Ισλανδό Υπουργό Αλίας στις 6 Ιουνίου την τελευταία φορά σας ενημέρωσα γιατί ήταν απόφαση που έλαβε και το Συμβούλιο το οποίο μου ζήτησε να πάω και να συζητήσω με τον Ισλανδό Υπουργό και ε, εγώ θεωρούσα ότι ήταν σημαντικό να δώσουμε μια ευκαιρία στην ε, νέα Ισλανδική κυβέρνηση να εκτιμήσει την κατάσταση και να αποφευχθεί η λήψη εμπορικών μέτρων. Δεν ε, μου έδωσαν μέχρι τώρα κανένα θετικό δείγμα ο Έδωσα οδηγίες λοιπόν να με πρόταση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση της Κομισιόν να ε, κατονομάσει τη χώρα ως χώρα που επιτρέπει την αναρχιαλία. Εν προκειμένου το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί ε, προσηκόντως ε, για κάθε στάδιο της διαδικασίας και ελπίζω ότι θα οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις πριν από τις θερινές διακοπές. Η νήσι που έχουν παρόμοια συμπεριφορά, όπως και οι Ισλανδοί στο Σκουμπρί, πρόκειται να αντιμετωπιστούν και εκείνοι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διαδικασία. Αυτά ως προς αυτό το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, περάσαμε από διαδικασία πολύ θετική μεταρρύθμιση της πολιτικής. Η πρόσφατη πολιτική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ε, θέτει πολύ σημαντικά, σημαντικές προσδοκίες για πιο βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική αλίας. Στο μεσοδιάστημα θα λάβω όλες τις πρωτοβουλίες για να διευκολύνω τη νέα συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πολιετή σχέδια. Το έχω συζητήσει και με τη Λιθουανική Προεδρία το θέμα αυτό και θα ε, έχω συντάξει και θα ε, στείλω στη Λιθουανική Προεδρία αύριο μία επιστολή όπου τους ζητώ σύμφωνα με τη δήλωση που υπογράψαμε των τριών θεσμικών οργάνων να προχωρήσουμε και να συστήσουμε αυτή την ειδική ομάδα υψηλού επίπεδου, task force, για να εξευρεθούν κάποιες ε, οριστικές τελεσίδικες λύσεις. Έχουμε κάποιες ιδέες ε, για να διευκολύνουμε τις ε, διαδικασίες αυτές. Χρειάζομαι όμως μία επιβεβαίωση από τη Λιθουανική Προεδρία ότι ε, συνεχίζουν και δίνουν συνέχεια στο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ και για την επιστολή που θα ε, αφορά τα management plans, τα σχέδια διαχείρισης. Μιλήσαμε και με τον Λιθουανό Υπουργό και το τονίσαμε αυτό το θέμα και παρακαλέσαμε και η ομάδα αυτή η ειδική, το Task Force να γίνει. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Υπουργός αυτός κάνει σοβαρές προσπάθειες για την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης γιατί ξέρει ότι αυτό θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και για την ελία και για τα ψάρια. Τώρα για τα δύο άλλα θέματα να ρωτήσω κάτι. Για την υδατοκαλλιέργεια καταρχήν είπατε ότι θα καταρτιστούν εθνικά σχέδια. Υπάρχει κάποια προθεσμία για αυτά, δηλαδή μέχρι πότε πρέπει αυτά να κατατεθούν. Και είπατε επίσης ότι θέλετε και αναμένετε μια ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό για την υδατοκαλλιέργεια, χωριστή. Διερωτώ από ποιον προϋπολογισμό και μετά θα ισχύει αυτό. Γιατί συζητήσαμε για τον προϋπολογισμό και δεν θυμάμαι στις συζητήσεις να μιλήσαμε για χωριστή γραμμή ε, προϋπολογισμού για την υδατοκαλλιέργεια. Τι θα πρέπει να ε, γίνει για να το συζητήσουμε και αυτό ως κοινοβούλιο. Τώρα για το σκουμπρί. Πολύ σύνθετο θέμα και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεταξύ Φερών, Νήσων και ε, Δανίας και οι τριβές ξεπερνούν την προβληματική του σκουμπριού καθ' αυτού. Είναι πολιτική πια η διένεξη στη Δανία, έτσι μου είπαν. Οπότε ερωτώ, τι σημαίνει η λήψη εμπορικών μέτρων. Εάν δηλαδή κινήσετε αυτή τη διαδικασία, τι συνέπειες θα έχει συγκεκριμένα και έχουν όντως εξαντληθεί όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτά δεν μπορούμε να τα ανεχόμαστε. Αλλά φαίνεται ότι τώρα είναι μεγάλο το πολιτικό πρόβλημα και η σύγκρουση και θα ήθελα να ξέρω τι σημαίνει ας πούμε, η συγκεκριμένη λήψη εμπορικών μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Λόβεν, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας και που κάνετε διάλογο μαζί μας για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του βασικού κανονισμού ε, της κοινή ελευτικής πολιτικής σε σχέση με τη υδατοκαλλιέργεια ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και σημαντικό ήταν επίσης ότι ε, θέλαμε να μειώσουμε την εξάρτηση σε ζωοτροφές για την ε, υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να το πάρουμε λοιπόν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αν θέλουμε δηλαδή να ε, αλλιεύουμε μόνο για ηχθιάλευρα, ε, για να έχουμε υδατοκαλλιέργειες, δεν έχει νόημα αυτό, δεν είναι ανάπτυξη. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας για την ανάπτυξη, γιατί ουσιαστικά πρέπει να αλλιεύσουμε 4-5 φορές παραπάνω από αυτά που ουσιαστικά παράγουμε στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Οπότε αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής υδατοκαλλιέργειας ότι πρέπει να μειώσουμε την ε, εξάρτησή μας ε, από τις θαλάσσιες ζωικές πρωτεΐνες. Σε σχέση τώρα με τη ε, διαμάχη μεταξύ των Φερών Ίσων και της Δανίας, είναι πράγματι μία ατυχής κατάσταση. Κάτι θα ήθελα να πω, το οποίο, του οποίου έλαβα γνώση από κάποιους συναδέλφους από το Σουηδικό Κοινοβούλιο και άλλων σκανδιναβικών ε, ε, κοινοβουλίων είναι το Συμβούλιο των ε, Βορείων Χωρών, το Nordic Council. Θέλει να υπάρξει μία λύση για το θέμα αυτό. Η άποψή τους για το όλο θέμα είναι, εντάξει θα δούμε διακυμάνσεις βεβαίως στα ε, αποθέματα οι οποίες θα επιμείνουν περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ε, αυτό είναι άλλωστε και το επιχείρημα ε, των φερών νήσων. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή και πώς τα ήχθη από θα ε, κινηθούν ειδικότερα τα άκρος μεταναστευτικά. Μπορεί να πάνε πολύ πιο βόρεια λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας στα ύδατα. Είναι λοιπόν ένα ευρύτερο θέμα το οποίο θα δημιουργεί όλο και περισσότερο συγκρούσεις ε, γιατί μοιραζόμαστε με τις ε, γειτονικέ μας χώρες τα ηχθιαποθέματα αυτά. Οι Φερόες Νήσι και ε, η Ισλανδία είναι γειτονικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που είπαν οι συνάδελφοι στο Βόρειο Συμβούλιο είναι να καθίσουμε και να συζητήσουμε για νέες παραμέτρους βάσει των οποίων να ε, διανέμουμε ε, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα ε, ή τις αλλιευτικές δυνατότητες. Όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν την Ισλανδία, που προτείνει η Ισλανδία και η Φερόες νήσι, ο χρόνος δηλαδή που ξοδεύει κανείς στις διάφορες ζώνες, αυτό θα ήταν βέβαια μια πρώτη ε, φάση εξέβρεση λύση να καθίσουμε δηλαδή επιστημονικά να δούμε πώ θα μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτά τα αποθέματα, γιατί προφανώ θα μοιραζόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν ανήκουν ούτε στην Ισλανδία, ούτε στι Φερόε Νίζου, ούτε στην Ιρλανδία, ούτε στη Σκοτία, ούτε σε κανέναν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, αν το έχετε ακούσει από τους συναδέλφους του ε, Βορείου ε, Συμβουλίου. Είναι τέλος πάντων μια ιδέα που πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στίβενσον, παρακαλώ, ο αντιπρόεδρός μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, που ήρθατε και πάλι να μας δείτε. Ε, εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα με τα, τη δράση που προτείνετε Θα ήθελα και εγώ να μάθω ακριβώς τι σημαίνει εμπορικές κυρώσεις. Μπορούμε να θέσουμε κυρώσεις ε, μόνο ε, για το ε, σκουμπρί, τέλο πάντων για τα αποθέματα τα οποία είναι το αντικείμενο, το μήλον της έριδος ή και όλα τα συνδεδεμένα αποθέματα. Και αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος Λόβεν πριν από λίγο, Έχουμε, έχουμε κάνει πάρα πολλές ατελείωτες διαπραγματεύσεις ε, με την Ισλανδία και τις Φερόες ε, ε, νήσους. Εγώ Είχα μάλιστα συχνά πολύ ζωντανές συζητήσεις, διαμάχες με πρωθυπουργού πολλές φορές ε, ότι για 16 εβδομάδες αλλιεύουν για το 1 τέταρτο του έτους ε, και αυτό βέβαια τους δίνουν τι δυνατότητε να παίρνουν τα 3 τέταρτα των εχθιαποθεμάτων. Ε, βάσει του, των πορισμάτων του ISIS αυτό είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι έχει πια περάσει, έχει παρέλθει ο καιρός των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών. Η δική του πρόταση ήταν... Ε, να διαπραγματευτούμε και αυτό δεν ε, δούλεψε. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να ε, τους επιβάλλουμε κάποιο είδους κύριο και θα ήθελα να ρωτήσω τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο στην πράξη. Ο κύριος Γκάλαγκερ. Εγώ να καλωσορίσω την Επίτροπο και να την ευχαριστήσω που ήρθε να μοιραστεί τις απόψεις της μαζί μας για πολλά θέματα, κατευθυντήριες γραμμές για την υδατοκαλλιέργεια, για παράδειγμα, που είναι πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Τώρα το θέμα είναι να υπάρξουν και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Η Ιρλανδία, η χώρα μου που τη βλέπω πρώτη, χρειάστηκε πολύ από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελικό, όχι της παραγωγής, αλλά της εμπορίας αυτών των ψαριών. Και υπάρχουν πολλοί άριθμοι τομεί. Ο Επίτροπο ανέφερε τη σημασία τη υγεία και τη ασφάλεια. Και προσθέτω κι εγώ ότι το προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όλοι θέλουμε να έχουμε ε, υδατοκαλλιέργεια, όχι ως βάρος όμως του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας, ε, πρόσφατα ε, μια μελέτη έδειξε ότι ε, στις περιοχές με υδατοκαλλιέργεια δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και μάλιστα αυτό προήλθε, αυτά είναι στοιχεία από το, το Θαλάσσιο Ινστιτούτο που το επισκεφθήκατε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Καλό είναι λοιπόν να, παρακολου... να υπάρχει παρακολούθηση των ε, παράκτιων κρατών για να κρυθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες και καλό είναι να κάνετε σύσταση στα τη μελη να έχουν μία υπηρεσία, μόνο απευθυντική όπως λέμε, αντί να πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο, ε, σε διάφορες υπηρεσίες, ε, να υπάρχει μία υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Οπότε το, μέσα σε 12 μήνες θα έχει στηθεί ε, το σύστημα, ενώ τώρα παίρνει χρόνια. Ξέρουμε ότι για να λυθεί το πρόβλημα στη, της ανεργίας ε, πρέπει να ε, ε, παίξει ρόλο ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος όμως δεν θα επενδύσει σε κανένα πρόγραμμα και έργο εκτός και αν κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα και χωρίς να παραβιάζονται οι υφιστάμενοι κανονισμοί ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που για διάφορους λόγους ε, κολλησιεργούν. Εδώ είναι ευκαιρία να προχωρήσουμε. Ε, η Προεδρία μας μίλησε για ανάπτυξη, μεγέθυνση, θέσεις εργασίας και βιωσιμότητα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και ε, κυρία Επίτροπε ελπίζω να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις εκεί. Τώρα για το σκουμπρί εγώ ήμουν πολύ επικριτικός γιατί έλεγα ότι έπρεπε από πριν να αναλάβουμε δράση. Και τώρα χαιρετίζω τα βήματα που ελήφθησαν και για την Ρέγκα αυτή την Άτλαντο-Νορβηγική που αυξήθηκε κατά 145% το μεριδιό του. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η μακροπρόθεσμα αυτή. Και οι άλλοι, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισλανδία, εμείωσαν το μεριδιό τους κατά 23% δρώντας με υπευθυνότητα. Είναι ώρα λοιπόν να αναλυθεί δράση και βεβαίως η δανική κυβέρνηση ε, που συμμετείχε με τους υπουργούς. Δεν με εκπλήσει αυτό. Καλό είναι όμως να δώσετε συνέχεια στο θέμα και να κινηθούν διαδικασίες σε μια εβδομάδα, όπως είπατε νομίζω. Ε, ρωτώ κι εγώ όπως ο Στουάν Στίβενσον τι σημαίνουν τα εργαλεία που έχετε, ότι μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις απέναντι στις εισαγωγές όλων των ειδών ψαριών και όχι μόνο της Ατλαντονορβηγικής Ρέγκας. Γιατί αν ε, γίνει το τελευταίο, αυτό τι κύρωση είναι. Θα, θα τιμωρηθεί ένα πολύ μικρό, θα τιμωρηθούν κατά πολύ μικρό ποσοστό. Ελπίζω να συμπεριληφθεί και το ε, σκουμπρί και ε, τα άλλα είδη. Εγώ πήγα στην Ισλανδία και αν ήμουν ε, βουλευτής στην Ισλανδία θα ήμουν υπέρ γιατί σημαίνει πολλά αυτό για εκείνους. Από 20.000 τόνους ανέβηκαν στις 130.000 τόνους κουμπριού. Είναι εισόδημα αυτό ε, και για τους Ελίσσα αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση γιατί σπράττουν φόρους από αυτά. Τους καταλαβαίνω από, εκείνους από την πλευρά τους. Εσείς πήγατε όμως εκεί, συναντήσατε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη εκείνοι. Οπότε μην περιμένετε άλλο από το απαραίτητο. Όταν θα είστε έτοιμοι και θα έχει ετοιμαστεί η κοινοποίηση για την Ισλανδία, θα έχουν ένα μήνα καιρό για να αντιδράσουν και μετά από τον μήνα εσείς θα ε, προχωρήσετε στη λήψη των, στην επιβολή των κυρώσεων. Γιατί πριν από 12 μήνες που πήγα στην Ισλανδία, μου είπαν ότι δεν γίνεται με τίποτε αυτό. δε ε, ε, και εγώ τους είχα πει ότι δεν θα σας επιτραπεί να γίνει αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, θα δούμε τι θα επιτύχουν οι κυρώσεις. Δεν είμαι πολύ ε, αισιόδοξο. Νομίζω ότι θα χαρούν δε ιδιαίτερα αν τα μέτρα, οι κυρώσεις αφορούν μόνο ε, ρέγγα και σκουμπρί. Γιατί αυτό δεν είναι κύρωση. Τώρα για τα πολυετή ε, σχέδια, ε, όπως είπα και πριν στον Λιθουανό Υπουργό, θα ήταν ε, μεγάλη αποτυχία της Επιτροπής μετά από πέντε χρόνια ανταλλαγών απόψεων ε, αν δεν ε, είχαμε σύντομα, δεν έχουμε σύντομα τα πολιετή σχέδια και το Task Force είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι ο Υπουργός μας ήταν ξεκάθαρο σήμερα ότι υποστηρίζει απόλυτα τη διαδικασία αυτή και μάλιστα ε, θέλει να διασφαλίσει ότι οι μέλη αυτής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν στην Task Force. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ρωμέβα, έχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω μία ερώτηση και εγώ μετά από τα σχόλια που ακούστηκαν Θα να αναφερθώ στην ε, λαθρέα ε, αλληλεία και στην άναρχη. και τη συμπερίληψη νέων κρατών στον κατάλογο. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι έχει γίνει, τι μπορεί να γίνει περαιτέρω για τον κατάλογο των χωρών αλλά και των σκαφών αν έχει γίνει κάποια δουλειά, κάποια κίνηση προς την αυτή σχετικά με την γκάλπ. Ευχαριστώ κύριε Τόμας. Oui, merci Monsieur le Président. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για το διάλογο που κάνετε μαζί μας ε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς σε σχέση με την ιδιατοκαλλιέργεια να αναφέρω το εξής, ότι όσο η, κοινή, η μεταρρυθμισμένη κοινή αλληλευτική πολιτική αποσαφήνισε τους περιορισμούς και το πλαίσιο μιας αηφόρου αλίας, ε, στην ιδατοκαλλιέργεια νομίζω ότι δεν μπήκαμε στην ουσία του θέματος του τι ακριβώς είναι, τι θα πρέπει να είναι ε, η αηφόρος ε, υδατοκαλλιέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφόρων ε, τμήματων υδατοκαλλιέργειας, για παράδειγμα φυκιών ή ψαριών, δεν είναι ακριβώς ίδιες οι συνθήκες και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε διάκριση στους τρεις τομείς, μεταξύ των τριών τομέων της υδατοκαλλιέργειας. Ε, υπάρχει βέβαια και το θέμα ε, ε, των ηχθιαλεύρων, των τροφών στην υδατοκαλλιέργεια που είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων κάπως δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των αλλιευτικών αποθεμάτων. Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα με τη συγκέντρωση ε, στην υδατοκαλλιέργεια και μιλάω κυρίως για τους ηχθείες γιατί το είδαμε ε, ότι το οικοσύστημα της Νορβηγίας ε, λόγω της συγκέντρωσης του Σολομού και της απόρριψής του καταστράφηκε εντελώς και ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε εύθραυστο οικοσύστημα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δίνουμε στα ψάρια διάφορα αντιβιωτικά Ε, για τις διάφορες αρρώστιες που μπορεί να έχουν ε, ε, λόγω του περιβάλλοντος τους. Νομίζω ότι είναι πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να τα δούμε λεπτομερέστερα. Και για το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω, για το σκουμπρί, θα ήθελα να πω ότι είναι προβλήματα γειτονία, αλλά είναι πολύ σημαντικά γιατί έχουν να κάνουν με τους αλευτικούς πόρους και έχουν να κάνουν ε, με τα θέματα ε, των προτεραιοτήτων που επίσης έχουμε θέσει στην κοινή αλευτική πολιτική. Και αν στον ίδιο χώρο, όπως κάνουμε σήμερα, τελικά ε, καταλήγουμε να μην μοιραζόμαστε τα ίδια κριτήρια ε, τα κριτήρια εκμετάλλευσης αυτών των πόρων. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ε, είναι αθέμητος πια ο ανταγωνισμός, υπάρχει σίγουρα στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, και προκύπτουν πάση περιπτώσει πάρα πολλά προβλήματα. Και όπως είπε και ο Πατ Κόπ Γκάλεγκερ, δύο λύσεις υπάρχουν, ε, κυρώσεις, αυτή είναι η πρώτη λύση, άμεσες κυρώσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει πολύ νόημα να το πούμε, να τις αναφέρουμε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή που θα, από τη στιγμή που θα ζητήσουμε τις κυρώσεις αυτές μέχρι να επιβληθούν θα υπάρξει κάποια χρονική διαφορά. Και δεύτερη περίπτωση, αν κατάλαβα καλά τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2014 πρέπει να διαπραγματευτούμε εκ νέου τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης αλίας με τις ε, χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισλανδία, Νορβηγία. Ε, και νομίζω ότι ίσως τότε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε την επιλογή των κυρώσεων πιο πριν. Αλλά τότε τουλάχιστον θα μπορούσαμε, ε, κατά τη γνώμη μου, να ε, δράσουμε γρήγορα ε, προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που έχουμε πάρει εδώ και πολύ καιρό. Εν πάση περιπτώσει αυτή η απειλή θα έπρεπε να τους κάνει να ξανασκεφτούν τα πράγματα, να ξανασκεφτούν αν έχουν καταλάβει καλά τους κανόνες του παιχνιδιού. Ετησίως ε, η Επιτροπή είναι αυτή που ρυθμίζει τη διαχείριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών αυτών χωρών που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Το 2014 το, το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και ίσως είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε και καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ με την ανησυχία που εξέφρασαν οι συνάδελφοι και δει αυτά που είπε η κυρία Ουρίκη Ρόλους, ε, δηλαδή πως υπάρχουν προγράμματα ιδιαίτερα φιλόδοξα, αλλά οι πόροι, τα κονδύλια Εάν θυρίζονται στο Ταμείο Αλίας, μιλάμε για ένα ταμείο το οποίο συνολικά μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο ταμείο. Μιλάμε άρα για λιγότερα χρήματα και περισσότερους στόχους, περισσότερη φιλοδοξία για τα προγράμματα. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερα σημασία είναι η ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων εχθικαλλιέργειας, ε, μια εχθικαλλιέργεια που ε, αντιμετωπίζει δυσκολίε ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προσδιοριστεί σε σχέση με την παράκτεια και την ραστεμική αλεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι εναλλακτική λύση στην υπερεκμετάλλευση σημαίνει μια δίαιτα υγιεινή στον κόσμο και στην Ευρώπη το οποίο μπορεί, να επιτευχθεί με την σωστή εκπαίδευση, σωστή κατάρτιση των παιδιών μας για μια υγιεινή δίαιτα όπως ε, αυτή της ε, κατανάλωσης αλλιευμάτων ε, και ειδικά των ρημών που από την παράκτη τώρα, το θέμα της ηχθειοκαλλιέργειας παρατήρησα ότι αναπτύσσεται με τρόπο διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή. Άρα οι εγγύησει ποιότητα ε, για τον ε, καταναλωτή διαφέρουν και ζητώ όλες οι χώρες που έχουν κάποιους κοινούς δείκτες ε, προκειμένου π.χ. χωρίς να αναφέρω κάποια χώρα να πω ότι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν ε, έχω κανένα πρόβλημα όταν ε, πρόκειται να ε, κάνω μια επιλογή σε θέματα αλλιευμάτων, δηλαδή π.χ. το λαβράκι. Το καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτό που τρώει, να γνωρίζει την ποιότητα, μετά από πόσες μέρες το καταναλώνει. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία προβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ε, λοιπόν, εσείς έχετε ένα πρόγραμμα εργασίας, ε, ε, έχετε τη θεματολογιό σας, αλλά υπάρχουν κάποια όρια που δεν εγγυώνται αυτή την ισορροπία και αυτή την ασφάλεια και διασφάλιση του καναλωτή. Και η ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι αυτή και αλλά και να λάβετε υπόψη σας ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν είναι πολλές φορές πολύ σοβαρότερα από αυτά που αναφέρθηκε εδώ, όπως ε, αυτά που αφορούν πρακτικές και είμαι της άποψης ότι για να εφαρμόσουμε κυρώσεις ε, και να τις επιβάλλουμε διότι η νομοθεσία πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Χρειάζεται όμως περισσότερη πόρη, περισσότερα κονδύλια για μια επιβολή για την επιβολή της νομοθεσίας. Τώρα, αν έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία, δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να την επιβάλλουμε, για να εφαρμόσουμε, τότε ο καθένας θα κάνει ό,τι του αρνητικά το δοκούν και η ερώτησή μου έχει ως εξή. Συμφωνώντας ότι θα πρέπει να επιτευχθούν η ισορροπία, πρέπει να έχουμε προγράμματα για μια καλλιέργεια που θα είναι βιώσιμη, και θα παρέχει εγγυήσεις ε, διατροφικές και όλα αυτά τα κονδύλια, τα απαραίτητα θα προκύψουν από αυτόν τον μικρό προϋπολογισμό, αυτό το μικρό ταμείο. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, ούτε το ταμείο πρόκειται να αποκτήσει ξαφνικά μερικά δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον. Ε, την περίοδο 2013-2020. Λίγα μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, ε, ε, μόλι ότι είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Θα πρέπει να αφήσουμε να καταπέσουν άλλα θέματα πολύ σημαντικά όπως οι απορρίψεις, η παράνομη αλληλεία, Νομίζω ότι η πρικοδότηση του Ταμείου είναι μικρή. Είναι πολύ λίγη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Να σας ρωτήσω και εγώ κυρία Επίτροπε. Αυτά σας καλωσόρισα προλίγου να σα πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Επιτροπή μετά από την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν όλοι, αλλά και η Κομισιόν για να καταλήξουν τη συμφωνία. Ήταν σημαντικά αυτά τα οποία έγιναν ε, και υπόθηκαν από πολλού ε, Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να συνεργαστούμε τούτου λεχθέντος ε, σχέση με τα προγράμματα Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία, με τον Λιθουανό Υπουργό και φαίνεται ότι είναι οφασισμένοι να προωθήσουν αυτά τα προγράμματα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτό και θέλαμε να ε, τεθεί σε λειτουργία αυτός ο, αυτή ομάδα. Και αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει τις εργασίες της ε, και υπάρχει βούληση να υπάρξει δηλαδή, απεμπλοκή σε ένα ζήτημα το οποίο έχει, υπάρχει, έχει προκύψει εμπλοκή και κάτι άλλο επειδή δεν θέλω να σας κορυδεύω θα ήθελα να σας ζητήσω τι γίνεται με τα προγράμματα. Υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά όπως αυτό τη συμφωνία με το Μαρόκο ε, Ξέρω ότι προβλέπεται ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Ε, θα μπορούσατε να μα ενημερώσετε έστω και εντάχει τι προοπτικέ, τι προσδοκίε σα, ε, αν μπορούμε να καλύψουμε μια τελική συμφωνία ή και την ε, ε, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Και ένα άλλο ζήτημα, αυτό της Μαυριτανίας, είναι γεγονός ότι ε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν αναφορικά με τη συμφωνία με τη Μαυριτανία και θα ήθελα να μάθω εάν η Επιτροπή, αν η Επίτροπος προτίθεται να προωθήσουν το ζήτημα πριν φτάσει στην Ολομέλεια και κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εξέλιξη, κάποια συμφωνία. Όπως είχε υποθεί, υπάρχει δυνατότητα να καταγγελθεί η συμφωνία ή δεδομένων των περιστάσεων δεν θα το πράξετε ή θα ζητήσετε την ε, σύγκληση με τη επιτροπής. Ποια είναι η άποψη λοιπόν τη Κομισιόν για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και πριν από τι τερνέ διακοπέ να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση σα προκειμένου και εμεί να υιοθετήσουμε την δική μα πριν από την ε, προηγούμενη ολομέλεια που θα συζητηθεί τώρα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Καταρχήν για την υδατοκαλλιέργεια. Η ιδέα είναι να πάρουμε σχέδια διαχειριστικά από τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του χρόνου ή το αργότερο θα πρέπει τα εθνικά σχέδια διαχείρισης να τα πάρουμε μαζί με τους φακέλους που θα έρθουν για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών, οπότε τρόπον την να η χρηματοδότηση συνδέεται με τα σχέδια διαχείρισης, γιατί θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι μιλάμε όπως είπαμε για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και προγράμματα υδατοκαλλιέργειας βιώσιμα και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα έργα, τα προγράμματα και όλες οι αιτήσει για χρηματοδότηση θα ευθυγραμμίζονται με την νομοθεσία της, Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, για την υγεία κλπ. Αυτή είναι η γενική ιδέα για το πώς θα εργαστούμε. Ε, κατάλαβα ότι έχετε κάποιες ανησυχίες για την υδατοκαλλιέργεια γενικότερα, ιδιαίτερα για τα σαρκοφάγα είδη. Σας θυμίζω ότι η μισή μας παραγωγή προέρχεται από στρακοειδή, όταν μιλάμε για υδατοκαλλιέργεια, και πρέπει να προσθέσουμε εδώ και την παραγωγή ειδών που δεν είναι σαρκοφάγα, όπως ο Κυπρίνος. Ε, έχουμε λοιπόν λάβει μελέτες που μπορούν να αποδείξουν ότι μεταξύ των άγριων ψαριών ε, μειώθηκαν ε, τα ποσοστά σολομού και πέστροφας και αναμένεται να, να συνεχιστεί η τάση. Για να το διευκολύνουμε αυτό θα δώσουμε και κάποια κίνητρα, χρηματοδοτικά εννοώ, στα έργα, στα προγράμματα που θα μας δώσουν ιδέες σχετικά με τη μείωση του προβλήματος. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι τώρα μετά την απαγόρευση της ε, ε ξανά στη θάλασσα, πώς μπορούμε να έχουμε ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα που τα χρειαζόμαστε για ζωοτροφή ε, στον κλάδο της ύδατο-καλλιέργειας από παραλίευματα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους τρόπους και έχουμε μάλιστα και κάποια καινοτόμα προγράμματα στην Ευρώπη μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα αν έχουμε χρόνο σχετικά με τη χρήση των παραλίευματων, των παρεπιπτόντων αλιευμάτων και έχουμε και ένα πολύ καλό ισπανικό πρόγραμμα εδώ που χρησιμοποιεί ό,τι μένει από την κατεργασία των ψαριών για να γίνουν τα χθιάλευρα. Οπότε μπορούμε να βρούμε τρόπους και καλού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί? Διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ευρώπη δεν είναι μεμονωμένη, ε, δεν είναι απομονωμένη. Είμαστε σε ένα ανοιχτό κόσμο, εισάγουμε πολλά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, οι πολίτες μας καταναλώνουν τα εισαγόμενα αυτά ήδη, κατά 60-70%. Δεν έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά κάπου εκεί είναι οι εισαγωγές και η κατανάλωση των ψαριών από υδατοκαλλιέργεια. Και από πού προέρχονται, από εδώ και από εκεί και η υδατοκαλλιέργεια αυξάνεται κατά 10% ε, ετησίως και η δικιά μας που είναι η καλύτερη είναι στη στασιμότητα. Πρέπει να την προωθήσουμε με ωραίο τρόπο και καλές μεθόδους και χρειάζεται βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Αυτό είναι στις κατευθυντήριες γραμμές μας, θα συνεργαστούμε, νομίζω και θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε και να είναι και βιώσιμη η παραγωγή. Αυτή είναι η ιδέα. Λοιπόν, τελειώνω με την υδατοκαλλιέργεια και πάω στο εμπορικό μέσο και τις εμπορικές κυρώσεις για να σας δώσω πρόσθετες πληροφορίες όπως ζητήσατε. Από τότε που ανέλαβα, κληρονόμησα αυτή την κατάσταση με τις παράκτιες συμφωνίες και συζητήσεις και το πρόβλημα με την Ισλανδία και τις Φερόες και τις, μονόπλευρες αποφάσεις τους. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω απόλυτα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρνήθηκε ποτέ ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το μερίδιό τους. Από τότε που ανέλαβα το συζητήσαμε και ίσως θα θυμάστε ότι το συζητήσαμε το θέμα και εδώ, σε αυτή την Επιτροπή. Ήρθα εδώ, σας ενημέρωσα σχετικά με το τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις, ότι θα αυξήσουμε την προσφορά που θα τους κάνουμε, θα συζητήσουμε μαζί τους, θα πάμε να τους πείσουμε, δεν καινούργια θέματα αυτά συζητούμε στα πλαίσια της παράκτιας συμφωνίας εδώ και τρία χρόνια. Τι έγινε λοιπόν. Εμείς αυξήσαμε τις προσφορές για το σκουμπρί. Μπορώ να σας πω ότι διπλασιάσαμε την αρχική μας προσφορά διπλασιασμός. Γιατί? Γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας όχι μόνο τα ιστορικά δεδομένα, αλλά και αυτά που είπαμε για την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά υπόλοιπα. Και τι έγινε μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισαν εκείνοι να θέσουν μονόπλευρα ποσοστώσεις. Και για τις Φερόες και τη Ρέγκα πρέπει να τονίσω και ότι είναι δύσκολο να το χειριστώ και πρέπει και εσείς να είστε ενήμεροι. Θέλω να πω ότι οι Φερόες εγκατέλειψαν την τράπεζα των διαπραγματεύσεων, σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήρθαν και όλες οι χώρες εκπροσωπούνται, η Νορβηγία, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαν εμείς δεν θα συζητήσουμε άλλο, χαίρετε, φεύγουμε και θέτουμε ποσοστώσεις, τις ορίζουμε μονόπλευρα. Οπότε δεν υπήρχε περιθώριο. Αφού ενημερώθηκαν ότι εμείς θα ε, ε, χρησιμοποιήσουμε το εμπορικό μέσο, υποδέχτηκα τους υπουργούς, τους δανούς, ε, χαιρέτησα τις προσπάθειές τους ε, να βρουν συμβιβαστική λύση. Εξήγησα ότι αυτό που περιμένουμε από τότε που αυξήσαμε την προσφορά είναι μια αντιπροσφορά. Να πούν και εκείνοι κάτι. Και δεν είπαν ποτέ τίποτε περίμενα πάρα πολύ. Πάρα πολύ περίμενα. Και θα θυμάστε ότι αυτή η Επιτροπή ήταν πολύ πιεστική. Εσείς είσαστε που με επικρίνατε γιατί καθυστερούσα, ίσως το θυμάστε. Εγώ ήθελα να εξαντλήσω κάθε περιθώριο διαπραγμάτευσης. Αυτό έγινε. Τώρα λοιπόν τους είπα, ακόμα και τώρα, τους είπα ότι πριν οριστικοποιηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δεν μπορώ να τη σταματήσω εγώ, αλλά υπάρχει χρόνο. Πριν οριστικοποιηθεί η διαδικασία, ελάτε σε εμά, ελάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αντιπροσφορά σα. Τι πιστεύετε, ποια πρόταση μπορεί να γίνει για να αρχίσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων και να συμβιβαστούμε. Και δεν ήρθαν. Λένε ότι θα μας μηνύσουν, θα προσφύγουν, μας απειλούν. Τι να σας πω, δεν θέλω να σχολιάσω. Σας εξηγώ όμως ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Κατόπιν τούτου αντιλαμβάνομαι και πρέπει όλοι να αντιληφθούν όλοι γύρω από αυτό το τραπέζι ότι η σύγκρουση αυτή έχει πολιτική διάσταση. Έχει. Έχει πολιτική διάσταση. Αναφέρομαι στην πολιτική της Δανίας, αναφέρομαι στη διεθνή μας διεθνή πολιτική. Αλλά τι να κάνουμε, γι' αυτό είμαστε άλλωστε και τόσο προσεκτικοί σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού μέσου. Τώρα, για τη ρέγγα η διαδικασία υπάρχει. Για τα συναφή είδη, ίσως ε, γνωρίζετε ότι το εμπορικό μέσον έχει αυτή την πρόβλεψη, ε, εργαζόμεθα πάνω σε αυτό και διερευνούμε όλες τις δυνατότητες. Δηλαδή η δυνατότητα να συμπεριληφθούν κι άλλα είδη, συναφή είδη, αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει. Πάω τώρα στο σκουμπρί. Ε, κάνω συζητήσεις με τη νέα Ισλανδική κυβέρνηση. Ε, βέβαια οι Φερόες ε, έφυγαν και από εκεί. Και από τις διαπραγματεύσεις για το σκουμπρί έφυγαν και από εκεί. Είπαν εμείς ε, θα αποφασίσουμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα. Για την Ισλανδία. Όπως είπαμε, διπλασιάσαμε την προσφορά για το σκουμπρί και περιμένουμε αυτούς τι θα πούν. Αυτοί τι θα πούν. Τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, όταν συζήτησα με τη νέα κυβέρνηση, του έδωσα τη δυνατότητα να έρθουν με αντιπροσφορά σε εμά και υπο, τους υποσχέθηκα ότι αν συνέβαινε αυτό θα γινόταν νέος γύρος διαπραγματεύσεως. Αρνήθηκαν όμως και μέχρι τώρα δεν είπαν τίποτα. Λένε, μιλάνε γενικά, λένε ότι θέλουν βιώσιμη αλληλεία, αλλά δεν λένε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε πάλι δεν υπάρχει περιθώριο για μένα. Τώρα τι κάνουμε λοιπόν. Έχουμε μία πρόταση και τη συζητάμε εσωτερικά. Αναφέρομαι τώρα στο σκουμπρί. Η πρόταση αυτή δεν είναι μόνο για την Ισλανδία αλλά και για τις Φερόες. Και η πρόταση αυτή, έχοντας κατά το θέμα των συναφών ε, ειδών, είναι κάτι που πρέπει να τα αποφασίσουμε. Ελπίζω, περιμένω, πιστεύω ότι η τελική απόφαση που θα ληφθεί από την Επιτροπή θα είναι πριν από τις θερινές διακοπές, οπότε μπορώ να σας πω ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί όπως πρέπει για το ζήτημα αυτό. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες εργαζόμεθα μαζί με την Νορβηγία. Είμαστε σε επαφή με τους Νορβηγούς συναδέλφους, την Νορβηγική κυβέρνηση και υπάρχει συμφωνία πάνω σε αυτό. Ε, τώρα θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πριν από το τέλος της ελιευτικής περίοδου. Δεν θέλουμε δηλαδή να εξαντληθεί ε, από την υπεραλίευση αυτή η αλληλευτική περίοδος, γιατί ναι, μπορεί να συζητήσουμε για τον επόμενο χρόνο, αλλά τότε μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά. Και πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να έρθουν τα νέα επιστημονικά πορίσματα, γιατί έχω κάποιες ενδείξεις ότι δεν θα είναι καλά. Δεν θα πω περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να περιμένω τον Οκτώβριο να έρθουν τα επιστημονικά πορίσματα. Γι' αυτό θέλουμε να επιταχύνουμε σε αυτή την ε, αλλιευτική περίοδο να κάνουμε κάτι πριν τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει θα ε, διαπραγματευτούμε. Φέτος του χρόνου θα συζητήσω με ε, τις συμφωνίες με Ισλανδία, Νορβηγία και με όλους, αλλά ελπίζω ότι μέχρι τότε θα ε, υπάρξουν κάποιες κινήσεις διευκολυντικές για τη συμφωνία από την πλευρά τους. Αυτό είναι ο στόχος μας, να υπάρξει συμφωνία. Και βεβαίως να αναγνωρίσουμε τις ιδέες και τα δικαιώματά τους, αλλά ε, σε βάση λογική και πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτά για το εμπορικό μέσο. Είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητη κατάσταση αυτή, ευαίσθητο τομέα. Παρακαλώ, αν έχετε ιδέες, ελάτε σε μένα τώρα. Γιατί έχω αντιληφθεί ότι κάποια μέλη ε, δείχνουν κάποια προθυμία. Αν ε, ισχύει αυτό, πείτε το διότι αργότερα θα είναι πολύ αργά. Τώρα, για τα πολυετή σχέδια μπορώ να καταλάβω τις ανησυχίες σας. Και συμφωνώ και εγώ ότι είναι κατεπήγον το θέμα. Σας θυμίζω ότι τώρα τρέχουν κάποια πολυετή προγράμματα, τα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί θα πιέσω πιέσω δεν είναι καλή λέξη. Θα κάνω το πάνω να πείσω τη Λιθουανική Προεδρία ότι πρέπει να συσταθεί αυτή η ειδική ομάδα, η Task Force και ελπίζω να συσταθεί πριν από τις θερινές διακοπές ε, επίσης. Ελπίζω. Η Λιθουανική Προεδρία έχει συμφωνήσει, αλλά από τη συμφωνία μέχρι την πράξη υπάρχει μια διαφορά. Όλοι πρέπει να δουλέψουν από κοινού για να έχουμε επιτεύγματα. Για την άναρχη λαθρέα παράνομη αλληλεία, Αιουγιού, δεν έχω να σας πω καινούργια πράγματα, ειδήσει, αλλά σας ενημερώνω για το χρονοδιάγραμμά μας. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα θα θυμάστε, έχουμε τρεις χώρες που έχουν μείνει από τον πρώτο κατάλογο και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ε, προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα σε αυτές. Ε, αυτές είναι οι χώρες που δεν συνεργάζονται δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, μέχρι το τέλος του χρόνου μπορώ να σας αναφέρω κάποιες χώρες ε, για τις οποίες θα έχουμε καινούργια κίτρινη κάρτα και αυτές είναι μεγαλύτερες χώρες. Αναφέρομαι στη δική σας κριτική ότι κυνηγάμε μόνο τα μικρά ψάρια. Όχι, κυνηγάμε και μεγάλα και θα δείτε μέχρι το τέλος του χρόνου τι κάνουμε. Επίσης, να σας πω ότι τον Οκτώβριο υπάρχει ε, πρόθεση να σας δώσουμε ειδήσει και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις για τα δικά μας κρατημέλη, γιατί έχουμε περιστατικά ε, παραβίασης της νομοθεσίας και από κράτη-μέλη και σχεδιάζομαι να κάνουμε τον Οκτώβριο σχετική, σχετικές ανακοινώσεις. Αυτά μπορώ να σας πω για την παράνομη αναρχέλεια. Για το Μαρόκο ξέρετε ότι θα υπάρξει νέος γύρω των διαπραγματεύσεων, ελπίζω τελικώς την επόμενη εβδομάδα. Ε, η προσδοκία μου είναι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, για να είμαι δεν νομίζω ότι μένουν πολλά να γίνουν από τη δική μας την πλευρά, γιατί τους ε, δώσαμε την καλύτερη προσφορά ε, και για τα οικονομικά θέματα πήρε τελική μορφή της συμφωνία. Λάβαμε υπόψη μας και αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο, δηλαδή σεβασμός διεθνούς δικαίου κλπ. Θα δούμε. Ελπίζω ότι θα πάει καλά. Για τη Μαυρετανία το βασικό πρόβλημα και η βασική ανησυχία μας σε σχέση με αυτήν την συμφωνία είναι το θέμα της κερδοφορίας. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δαπανηθούν καλά τα χρήματα των φορολογουμένων Μέχρι τον προηγούμενο μήνα το επίπεδο αξιοποίησης αυτού του μέσου με βάση τις άδειες ε, προστιθέμενη αξία και αλλιεύματα είναι πολύ χαμηλά, οπότε σκεφτόμαστε αν είναι κερδοφόρος αυτή, επικερδής αυτή η συμφωνία. Από τότε όμως έχουμε κι άλλα, αποκτήσαμε κι άλλα στοιχεία. Αυξήσαμε τις άδειες πρόσφατα, έχουμε 11 άδειε στα πελάγια ήδη και κάποιες αφορούν μεγάλα σκάφη. Τα λιεύματα είναι ικανοποιητικά. Ελπίζω ότι όλη η ποσόστοση θα ε, ολοκληρωθεί στα πελάγια ήδη μέχρι το τέλος του έτους. Για τις γαρίδες δεν έχουμε ε, νέα. Για να συντομεύω, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η συμφωνία είναι καλή, αλλά ε, να πόκειται στα κράτη-μέλη και τους στόλους μας να τη δεχτούν ή όχι. Πρέπει να ελέγξουμε το θέμα της ε, κερδοφορίας και θα σας ενημερώσω στις αρχές του φθινοπόρου σχετικά με το τι θα κάνουμε. Αν υπάρχει κερδοφορία δεν έχω άλλο πρόβλημα. Το μόνο μου πρόβλημα είναι αυτό, αν αξίζει τον κόπο. Και όπως ξέρετε υπάρχει μια ρήτρα στη συμφωνία ότι αν τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιήσουν τις προσθέσεις δεν θα πληρώσουμε. Οπότε τα χρήματα των φορολογουμένων είναι εξασφαλισμένα εν πάση περιπτώσει. Αυτά και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε ο κ. Γκάλαχερ για μια σύντομη παρέμβαση. Με προκάλεσε να απαντήσω. Μας είπατε, η Επιτρόπος μας είπατε ότι αν θέλετε να μου πείτε κάτι, πείτε μου το τώρα. Έχουμε εξαντληθεί. Σας δώσαμε ένα ε, εργαλείο. Έχουμε περάσει τη φάση των ιδεών. Σε πρακτικούς όρους, να σας πω, είπατε ότι ελπίζετε να ισχύσει μέχρι το τέλος της, ε, του μηνός πριν ε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ σας σέβομαι, κύριε ε, πίτροπε. ε, όμως οι Ισλανδοί και οι νήσοι Φερόες είναι πιο έξυπνοι από εμά αυτή τη στιγμή θα περάσει ο χρόνο και θα πούνε ξεγελάσαμε μία ακόμη φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πάμε στην επόμενη χρονιά και όταν ε, ε, θα γραφτεί η ιστορία αυτής της θητείας θα πούμε ότι αποτύχαμε, γιατί είμαστε εδώ να προστατεύσουμε και ουσιαστικά μειώνουμε συνεχώς την αηφορία της αλληλείας. Θα είμαστε υπεύθυνοι για την εξάντληση των αποθεμάτων του σκουμπριού και είναι στο χέρι σας κυρία Επίτροπε να λάβετε γρήγορα μια απόφαση γιατί αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία νέο ε, κοινοβούλιο, νέο Νέα επιτροπή σημαίνει νέο παιχνίδι για τις Φερόες νήσους. Ε, βεβαίως είναι πολιτικός ευαίσθητο αυτό το θέμα, αλλά η ευθύνη σας είναι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό που σας λέω λοιπόν κυρία Επίτροπε, παρακαλώ να είστε γρήγοροι, να λάβετε δράση γρήγορη, γιατί αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα για το σκουμπρί, αν δεν υπάρξουν οι κυρώσεις, ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτε. Ε, είναι γραμμένο μέσα στο εργαλείο. Πρέπει να συμπεριληφθεί, διότι διαφορετικά, και αυτό θα είναι το τελευταίο που θα πω, αν ήταν μόνο το αν δεν κάνουμε τίποτα για το σκουμπρί, δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτε άλλο. Αν κάνουμε κάτι για το σκουμπρί, τότε και τα συναφή ήδη συμπεριλαμβάνονται. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για να κλείσει Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που είπε ο κύριος Γκάλαχερ. Βεβαίως, να το λάβω υπόψη και αυτό. Είμαι υποχρεωμένη να λάβω υπόψη όλες τις απόψεις ε, όλων των ε, μελών της Επιτροπής. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που βρεθήκατε ανάμεσά μας. Είμαστε στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια. Bien, continuamos con el punto número 10. Συνεχίζουμε με το σημείο 10 της Μεσαίας Διατάξεως, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014, ε, τμήμα 3. Η Κομισιόν στις 26 Ιουνίου δημοσίευσε τον προϋπολογισμό της, όπως γνωρίζετε, κάτι το οποίο μας ε, εμπόδισε το να έχουμε μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Σήμερα ο εισηγητής κ. Ριμπελίνη θα μας ε, μιλήσει για τι ε, προτάσει του, τι συστάσεις του, αλλά προηγούμενα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, ώστε να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού τη ε, Κομισιόν. Και μετά θα λάβει το λόγο κ. Βελίνη και οι υπόλοιποι βουλευτέ ε, που θα θελήσουν να ομιλήσουν. Thank you, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Η Κομισιόν ε, ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού 26 Ιουνίου αργότερα, όπως είπατε, από ό,τι άλλες χρονιές, για γνωστούς λόγους σε όλους, λόγω των συζητήσεων για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρά την καθυστέρηση θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η συνθήκη. Αυτό που σημαίνει είναι ότι επειδή ε, ήταν μεθύστερο το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρουμε ακόμα τη θέση ε, του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού. Υπάρχουν λίγα πράγματα που είναι σίγουρα. Ένα σίγουρο είναι ότι σίγουρα θα υπάρξουν προτάσεις για περικοπές από το Συμβούλιο στις προτάσεις μας, γιατί η πείρα δείχνει ότι αναπόφευκτα πάντα αυτό συμβαίνει. Τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί στην αρχή, είμαστε στην αρχή της νέας προγραμματικής περίοδου. Αν και δεν έκλεισε η συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ακόμα. Ξέρουμε ότι οι συζητήσεις ε, που έγιναν τέλος Ιουνίου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό και μόνο η νομική πράξη πρέπει να εγκριθεί το φθινόπωρο όταν το Κοινοβούλιο θα έχει επαρκή διασφάλιση σχετικά με την διαθεσιμότητα των υποχρεώσεων πληρωμών για το 2013 και το άλλο κομμάτι του προϋπολογισμού θα έχει εγκριθεί. Οι προτάσεις που υποβάλαμε εμείς για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλληλεία συνάδουν απόλυτα με τη συμφωνία ε, του τέλους Ιουνίου που εγκρίθηκε ε, την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Τώρα, Πού βρισκόμαστε στον προϋπολογισμό. Το ποσό που προτάθηκε στις υποχρεώσεις για το 2014, αυτή είναι η συνολική εικόνα για όλο τον προϋπολογισμό, είναι 142,5 δις ευρώ. Και το ποσό που προτείνεται για τις πιστώσεις πληρωμών είναι 136 δις ευρώ. Τώρα, τι αντιπροσωπεύει αυτό όταν εκφραστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ένωσης για το 2014. Οι υποχρεώσεις είναι 1,75% και οι πληρωμές είναι 1,01%. Υπάρχει μια σημαντική καινοτομία στον προϋπολογισμό φέτος, ότι δηλαδή η Κομισιόν έκανε επίμονη προσπάθεια για απλούστευση. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση του αριθμού των γραμμών του προϋπολογισμού και νέο τρόπο παρουσίασης των ε, εγγράφων. Κάθε τίτλος είχε με ένα αριθμό δραστηριοτήτων μέχρι τώρα και στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλλιές είχαμε 7 δραστηριότητες επιχειρησιακές. Τώρα, τώρα αυτό ήταν έδινε μια κάπως αποσπασματική εικόνα Στι δαπάνε στο τομέα αυτό τη πολιτική που δεν τα παρουσιάζει όλα μαζί. Η Κομισιόν προτείνει προπολογισμό για όλου του τομεί πολιτική, όχι μόνο για θαλάσσιες υποθέσει και αιλία, που στηρίζεται σε αυτές τις ε, δηλώσει προγραμματικέ, Μειώνονται λοιπόν τα κεφάλαια, απλουστεύονται στον προπολογισμό και σε ό,τι αφορά τι θαλάσσιες υποθέσει και την αιλία πάμε σε δύο προγραμματικέ δηλώσει. Μία προγραμματική δήλωση ανταποκρίνεται στο Ταμείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αιλίας και το άλλο αναφέρεται στο διεθνές κεφάλαιο. Οπότε αν δούμε τι έχουμε σε αυτούς τους τομείς, στην πρόταση MMF έχουμε επιμερισμένη και άμεση ε, διαχείριση. Οι περισσότερες δαπάνες είναι στην επιμερισμένη. Και ως μέρος των προτάσεων, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε οι δαπάνες που ήταν στην άμεση ε, διαχείριση να πάει στην ε, επιμερισμένη, γιατί πιστεύουμε ότι καλύτερα θα εκτελεστεί ο προπολογισμό έτσι και θα δώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε κάποιες ροές από τον προπολογισμό στα κράτη-μέλη. Στην επιμερισμένη, λοιπόν, θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και υδατοκαλλιέργεια και αλληλεία Θέλουμε ε, υποχρεωτικές ε, δαπάνες, δαπάνες για συλλογή δεδομένων, αντισταθμιστικά μέτρα για τις ε, απομακρυσμένες περιοχές και το, την αποθεματοποίηση η οποία τώρα σιγά σιγά εξαλείφεται. Τώρα έχουμε στο δεύτερο κομμάτι πάλι δαπάνες ε, για τον έλεγχο και εδώ κοιτάμε ε, επιμερισμένο έλεγχο και ε, επιθεωρήσεις από τους επιθεωρητές της Ένωσης. Επίσης δαπάνες σε σχέση με το παρατηρητήριο της αγοράς που έκανε και έκθεση θαλασσινών πριν από λίγους μήνες. Επίσης δαπάνες για επιστημονικά δεδομένα που επηρεάζουν τις πολιτικές και τις αποφάσεις. Δαπάνες για τη διακυβέρνηση ε, δηλαδή τα γνωμοδοτικά συμβούλια κυρίως εννοούμε εδώ και δαπάνες για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τέλος τις προαιρετικές εισφορές που γίνονται στις ε, περιφερειακές οργανώσεις των αλλιέων. Τώρα, στον άλλο τομέα που χρηματοδοτείται εκτός αυτού του EMFF που έχουμε το διεθνές κεφάλαιο, εδώ έχουμε προγραμματική δηλήρωση, έχουμε τις, προ... τις υποχρεωτικές εισφορές που καταβάλλονται σε αιτήσια βάση και όλες τις πιστώσεις για την υποστήριξη των ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης για την αλληλεία, ε, τέλη πρόσβασης κλπ. Και εκτός πεδίου εφαρμογής του EMFF έχουμε και ε, συνεισφορές στην υπηρεσία ελέγχου αλληλείας. Δύο λόγια για τα ποσά τώρα σε κάθε τομέα. Τώρα για το EMFF, το Ταμείο, 84% προτείνεται για αυτό στον τομέα της πολιτικής. Τώρα για το ποσό ε, στις υποχρεώσεις μιλάμε για 1 δις 63 εκατομμύρια ευρώ και στις πληρωμές μιλάμε για 813 εκατομμύρια ευρώ. Για το ταμείο, το EMFF, ε, έχουμε πολλές πληρωμές που ουσιαστικά είναι για τα υφιστάμενα προγράμματα από την τωρινή περίοδο, γιατί του χρόνου μιλάμε για προκαταβολές που θα πληρωθούν στα κράτη-μέλη, περίπου 85% των πληρωμών που απαιτούνται για το Ταμείο ε, θα αφορούν τις ε, εκρεμείς υποχρεώσεις. Τώρα στην επιμερισμένη διαχείριση έχουμε 85% που καλύπτει τις, ε, τους τομείς που ανέφερα πριν. Στην άμεση διαχείριση έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, λίγο παραπάνω από 100 εκατομμύρια στο Ταμείο που θα καλύψουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, μέτρα εφαρμογής, ελέγχου, επιστημονικά πορίσματα και γνώσεις. Επίσης έχουμε κάποια συνοδευτικά μέτρα για την κοινή ερευνητική πολιτική, έχουμε μελέτες, επιστημονικά πορίσματα, ε, έλεγχο και επιβολή, ε, διεθνείς οργανισμούς, ε, υποχρεωτικές εισφορές ε, για τη θαλάσσια πολιτική. Πώς θα μοιραστούν αυτά τα 100 εκατομμύρια, 43 για τη θαλάσσια πολιτική και 60 για τα συνοδευτικά μέτρα. Τέλος, για το, την υπηρεσία ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλίας. Ένα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως ξέρετε, ήταν ότι όλες οι υπηρεσίες, οι φορείς, οι οργανώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στη μείωση του προσωπικού, οπότε έχουμε περικοπή μέσα σε πέντε χρόνια για την Κομισιόν 1% και όλα τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες. Οπότε το EFCA, EFSA, ε, εδώ είναι το προπολογισμό στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν το 2013 και τέλος, η e Και τέλος να πω δύο λόγια για τη διεθνή αλληλεία. Εδώ έχουμε 14% των πιστώσεών μας ως επιτοπλίστων για τις ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες εταιρικής σχέσης. Ένα μικρό ποσό είναι για ε, υποχρεωτικές ε, εισφορές για τους οργανισμούς των αλλιέων. Εδώ είναι ο ίδιος ο προϋπολογισμός το 2013 και το 2014. Οι περισσότερες πιστώσεις για τις συμφωνίες αλλιέας είναι στο αποθεματικό και έτσι πρέπει γιατί η νομική βάση επί της οποίας θα δράσουμε δεν έχει ακόμη εγκριθεί και αν δεν ισχύει ε, η νομική βάση την 1η Ιανουαρίου, τότε οι πιστώσεις θα πρέπει να μπουν στο αποθεματικό. Για τις υποχρεωτικές φορές ε, στους οργανισμούς αλλιές είναι ένα μικρό το ποσό, αλλά έχουμε μια αύξηση εκεί, διότι προβλέπουμε νέες συστάσεις τέτοιων οργανισμών που θα ολοκληρωθούν το 2013 και θα πρέπει και αυτούς να τους καλύψουμε ε, συμπεραίνω είναι σημαντικό ο προπολογισμό μα, ο πρώτο στη νέα προγραμματική περίοδο, η πιστό στα συμπεράσματα ε, για το Ταμείο, είναι καινοτόμο με την έννοια ότι έχουμε κάνει απλουστεύσει και είναι και καινοτόμο ε, υπό την έννοια ότι περνάμε από την άμεση στην επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señor Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν που μας έδωσε χρήσιμες προφορίες διότι το σχέδιο γνωμοδότησης που είχα ήδη ετοιμάσει πριν μερικές εβδομάδες δυστυχώ ε, δεν είναι πλήρης δεδομένου που ότι δεν έχω λάβει ακόμα το σχέδιο προπολογισμού 2014 διότι όπως δήλωσε και η Κομισιόν δημοσιεύθηκε την 26 η Ιουνίου. Φυσικά εγώ δεν παρετούμε από το να κάνουμε μια παρουσίαση ως εισηγητής της Επιτροπής Αλίας για τον Προπολογισμό 2014 και να δώσω κάποιες πληροφορίες στους συναδέλφους. Πιστεύω πως θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα πέντε σημεία που εγώ θα παρουσιάσω ως τροπολογία στο σχέδιο γνωμοδότησης που ήδη λάβατε και αναγνώσατε. Το πρώτο σημείο είναι ότι εκτιμώ θετικά τον τρόπο αλλαγής της διαχείρισης ε, από τον έμεσο στον επιμερισμένο που στηρίζει τη δαπάνη των κρατομελών στο θέμα της, του ελέγχου και της συλλογή στοιχείων. Νομίζω πως αυτή η αλλαγή μπορεί να διευκολύνει ε, τα κράτη-μέλη, την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, συγγνώμη, και την άλυψη των δεσμεύσεών τους, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ορθή ε, εφαρμογή της ε, αλληλευτικής πολιτικής. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ενημερώθηκε ότι σημαντικά ποσά σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, με τρίτες χώρες για μια φόρο αλληλεία αποκλείστηκαν παραμέληθηκαν και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Δηλαδή ποια είναι ε, τα ποσά, τα ακριβή ποσά που ε, τέθησαν ε, κατά μέρο και καλό την Κομισιόν να συνεχίσει να, τις προσπάθειες της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες προκειμένου να ε, υλοποιηθούν σύντομα οι συμφωνίες για τον τομέα της αλίας ε, με τρόπο επωφελή για όλους και να χορηγηθούν τα πρέτα κονδύλια στον προπολογισμό προκειμένου ο Ευρωπαϊκός Στόλος ε, να επωφεληθεί τα μάλλον την περίοδο του 2014, την ελευθερική περίοδο. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι οι ε, περισσότερες ε, καταβολές ε, για πληρωμές του 2014 θα καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος 2007-2013 και αυτές οι πληρωμές είναι απαραίτητες για να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις που λάβαμε στο παρελθόν. Τέταρτον, θα πρέπει να πληροφορήσει το Συμβούλιο και να το ειδοποιήσει ότι θα πρέπει να μην κάνει περικοπές στον προβλησμό διευθύνει 14 Αυτές οι περικοπές θα έχουν τραγικές συνέπειες ε, πρώτο έτος εφαρμογής του νέου προγράμματος που ενεργοποιήθηκε για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγέ ε, σύμφωνα με τους στόχους της ε, Προγράμματος Ευρώπη 2020. Και τέλος, νομίζω ότι ο του 2014 θα πρέπει να συνοδεύει με τρόπο αποτελεσματικό την κοινή αλληλευτική πολιτική και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που μεταρρυθμίστηκαν προσφάτως. Να καταλήξω τονίζοντας την σημασία που έχουν τα, προγράμματα, τα πιλωτικά προγράμματα που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου με τις ευκαιρίες να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιστοπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ε, για την εφαρμογή αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων και να παρουσιάσει το των δυνατών τα πρώτα αποτελέσματα και τις σχετικές εκτιμήσεις. Φυσικά βασίζομαι στην συνεργασία όλων των συναδέλφων της Επιτροπής Αλίας και για υποβολή τροπολογιών στην ε, νομοδότησή μου προκειμένου να συμμετέχουμε όλοι στην διαδικασία λοιπόν του προβλήμου 2014, μολονότι αντιμετωπίζει με περίοδο κρίσης, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ε, Ευρωπαίων αλλήλων και των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Βέννη, κύριε Φράγκα. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε με τα στοιχεία που έχουμε για τον προβλησμό που είναι κατακαιρματισμένα, ελληπή κλπ. Και η ανάγνωση του Συμβουλίου δεν έχει δημοσιευθεί στο τέχος που περιλαμβάνονται οι νομικές βάσεις κλπ. κλπ. Θα ήθελα σε αυτού να ζητήσω από την Κομισιόν το 11.666. Αυτή είναι μια γραμμή απλούρα ΦΕΠ που θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να το γνωρίζω. Στο δεύτερο, το ζήτημα τη ε, υπηρεσία ελέγχου. Πιστεύω ότι υπάρχουν περικοπές για τις υπηρεσίες γενικότερα και δεν θα πρέπει να γίνουν ε, παντού στι περικοπέ, αυτό είναι άλλο ζήτημα τώρα για την προπαρασκευαστική δράτη, το Monitoring Center ε, for Fishing Prices που αναφέρεται ως PM είναι κάτι το οποίο δήλωσε η Επίτροπο φέτος. Γιατί υπάρχει μόνο PM προβεμόρια, δεν προβλέπεται κάποιο προπολογισμό, κάποια ποσά, ούτε δεσμεύσει ούτε πληρωμές αυτό είναι ένα ζήτημα που, το οποίο φέτο έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα, έγινε παρουσίαση από επιτρόπου και βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα με πρικοδότηση, μόνο ένα προσυπόμνηση PM. Αυτά προ το παρόν θα πρέπει να μελετήσω σε βάθο ε, τις αλλαγέ που έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει πολλές. Α, και κάτι ακόμα, το λέω και προ τον εισηγητή. Φαντάζομαι κύριε εισηγητά πως εσείς ε, όταν θα έχουμε το σχέδιο προπολισμού και φυσικά θα ε, γνωρίσουμε τις ε, γραμμές, ε, θα επανυποβληθεί το σχέδιο προπολισμού ως ελάχιστο, ως, ως κατελάχιστον. Εντάξει. Είναι καταφαντικά ο εισηγητής. Κυρία Λέβεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Ε, δεν έχουμε δει αριθμητικά στοιχεία ακόμη. αλλά αν δούμε τα έγγραφα συνεδρίαση στο φάκελό μας ε, ή στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει σχέδιο έκθεσης ε, δικό σας κύριε Ριβελίνη, οπότε δεν μπόρεσα να διαβάσω τίποτα και είναι λίγο δύσκολο να σχολιάσω συνεπώς. Μια ανόητη ερώτηση σε σχέση με την Συμφωνία εταιρική σχέση για την αηφόρο αλληλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι εκτός ε, του IMFF. Ε, ε, ποιο, τι ποσό ακριβώς, τι ποσό προβλέπετε, ποιο είναι το ύψος του ποσού σε σχέση με, τις υποχρεωτικές, με την υποχρεωτική συνεισφορά των περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλίας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ε, ναι, καταλαβαίνω, δεν έχετε έγγραφα και σας καταλαβαίνω, εγώ έχω τα έγγραφα και πάλι περίπλοκο το βρίσκω, οπότε καταλαβαίνω το πρόβλημά σας. Οποιαδήποτε μετάβαση, αλλαγή από το ένα σύστημα παρουσίασης ε, προϋπολογισμού σε άλλο σύστημα παρουσίασης προϋπολογισμού Παίρνει κάποιο χρόνο ε, να προσαρμοστεί κανείς αυτό και βεβαίω ευχαρίστως να σας εξηγήσουμε ό,τι χρειάζεστε, είτε δημερό είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως θέλετε. Ευχαριστώ να το κάνουμε αυτό. Αυτό είπε η κυρία Φράγκα, είναι δύσκολο να δει κανείς ε, τις αλλαγέ. Προσπαθήσαμε να δείξουμε στο έγγραφο του προπολογισμού τις αλλαγές, πώς μία γραμμή έχει συγχωνευτεί με μία άλλη ε, ή αν κάποια έχει αλλάξει τίτλο κλπ. Όσον αφορά τώρα τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Φράγκα, για την 11.06.60 ε, γραμμή και το ερώτημα ήταν ε, αν ε, είναι υποχρεώσεις ε, που θα τις διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, αυτές είναι κοινή διαχείρισης. Είναι όλες οι επιστώσεις υποχρεώσεων που θα έχουν στην επιμερισμένη διαχείριση στα κράτη-μέλη, φόρο, υδατοκαλλιέργεια, φόρο αλία, συλλογή δεδομένων, όπως επίσης ε, και για τις άκρως απόκεντες περιοχές, τα προγράμματα. Αν θέλετε να, να, για να σας το παρουσιάσω, είναι σαν EFF+, σαν Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας Plus υπάρχει για τον ε, οργανισμό, την υπηρεσία ελέγχου μια διαφορετική ε, ξεχωριστή γραμμή, η 64 και είπα, όπως, ε, όπως είπα τα επίπεδα είναι ίδια με τις περασμένες χρονιάς και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι διαφορετικά τα ποσά. Υπάρχει μια εξήγηση. Όταν μια υπηρεσία υποεκτελεί τον προϋπολογισμό της και όλες οι υπηρεσίες το κάνουν αυτό, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης του υπολοιπόμενου ποσού και αυτό το ε, μη εκτελεσθέν ποσό επιστρέφει στην υπηρεσία τελικά. Όταν λοιπόν υπολογίζουμε τον προϋπολογισμό, βλέπουμε πού βρισκόταν, βρισκόταν το 2013. Ξέρουμε το επίπεδο ε, πλεονάσματος από την ε, περασμένη χρονιά. Μειώνουμε λοιπόν το πλεόνασμα και το το ποσό που προτείνουμε είναι το ποσό ε, που τους επιτρέπει να επανέλθουν στο επίπεδο του 2013 αν συμπεριλάβουν το πλεόνασμα. Όσον αφορά τώρα τις εταιρικές συμφωνίες αηφόρου αλίας, τα συνολικά ποσά 145 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 145 σε ε, υποχρεώσεις. Ε, σε υποχρεώσεις και σε πληρωμές είναι το ίδιο ποσό. Ε, για τις εταιρικές συμφωνίες που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου ε, του 2014 είναι 22,3 εκατομμύρια ε, και για το αποθεματικό, και αυτό το λέω για αυτό που ρώτησε ο κύριος Ριβελίνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες λαμβάνονται υπόψη, ότι υπάρχουν αλλιευτικές δυνατότητες υπό τις συμφωνίες αυτές ε, το συντομότερο δυνατόν και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, ότι θα συμβεί αυτό. 122,6 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ποσό. Όταν λέω ότι είναι εντός ε, του Ταμείου Αλίας. Ε, ο λόγος είναι απλός. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη νομική τάξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχουμε μια βασική νομική πράξη που μας δίνει τη δυνατότητα να ε, εκταμιεύουμε τα λεφτά. Και το ε, Ταμείο μας δίνει αυτή τη βάση, όμως με τις εταιρικές συμφωνίες η νομική πράξη, η βασική πράξη είναι η απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας που δίνει τη σύμφωνη γνώμη σε αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα ουσιαστικά θα είναι αλληλοεπικάλυψη το να τα έχουμε και τα δύο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας αλλά και στην απόφαση του Συμβουλίου ε, που θεωρείται η βάση μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Τώρα, όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, προγράμματα πάρει προς τον κύριο Λιβερίνη. ε, θα σας ενημερώσουμε για το τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε και θα σας ενημερώσουμε βέβαια και τα, για τα αποτελέσματα της δουλειάς ως σήμερα. Για να ολοκληρώσουμε το ερώτημα που έθεσε η κυρία Φράγκα σε σχέση με την EU ε, MAFA, ε, Η δημοσιονομική γραμμή είναι 11.06.62.05. Πρόκειται για ένα, ευρωπαϊκό, για ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκών αγορών 4.405 ε, εκατομμύρια ε, είναι οι πιστώσεις υποχρεώσεων και 2,2 οι πιστώσεις πληρωμών. Ο κύριος Ριβελίνη για να κλείσουμε τη συζήτηση. Είχα παρουσιάσει ένα αρχικό σχέδιο που βρίσκεται στον φάκελο, αλλά επειδή δεν είχα τα στοιχεία, τους αριθμούς δεν μπορούσα παρά να παρουσιάσω αυτό το σχέδιο το γενικό. Θα περιμένουν λοιπόν τα στοιχεία. Ακούσαμε από την Κομισιόν ε, κάποια θέματα. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα ότι φυσικά θα πρέπει να αγωνιστούμε ώστε τα ποσά να είναι τουλάχιστον αυτά των προηγουμένων ετών. Γι' αυτό καλό την Επιτροπή να μην κοιτάξει μόνο τα πλεονάσματα και να αφαιρέσει αυτά τα πλεονάσματα, αλλά και εκεί όπου δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και υπάρχουν δυσκολίε να φροντίσει να τα εξισορροπήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ό,τι αφορά τα ποσά και τα σπόρους όπως είπε η κυρία Φράγκα, η κυρία Λεβίν να μπορέσουμε να βρεθούμε στο ύψος των προηγούμενων ετών. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη να πω σε όλους ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών τόσο για το σχέδιο νομοδότησης όσο και για το τμήμα του προπολογισμού ε, είναι η 12, 12 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. 12 Ιουλίου. Επίσης υπάρχει δυνατότητα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ή 40 βουλευτέ να υποβάλουν τροπολογίε ε, επί του προβλησμού μέχρι το μεσημέρι τη 5η Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, 12.00. Χρειάζεται η Επιτροπή Συνολότη ή 40 βουλευτέ μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου. Δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, αλλά η ανάγνωση του Συμβουλίου είναι τα τέλη Ιουλίου. Πώς μπορούμε να καλυθέσουμε τροπολογίες εμείς επί των ποσών, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με την ανάγνωση του Συμβουλίου. Λοιπόν, η ημερομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου, εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μία Επιτροπή Κοινοβουλευτική ή 40 βουλευτές, διότι είναι αδύνατον. Δεν μπορούμε να εκπλώσουμε αυτή την υποχρέωση. Εμένα το ίδιο μου κάνει έτσι κι αλλιώς, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταθέσω μια τροπολογία στο όνομά μου αν δεν έχω την υποστήριξη της όλης επιτροπής ή 40 βουλευτών. Και εγώ δεν μπορώ να την καταθέσω διότι δεν, η ε, ολοκλήρωση του Συμβουλίου γίνεται στα τέλη του Ιουλίου. Θα ζητήσω λοιπόν τις τεχνικές ε, ε, από τις τεχνικές υπηρεσίες τι συμβαίνει. Θα πρέπει να είναι η Επιτροπή στο σύνολό τη ή οι 40 βουλευτές, διότι δεν προβλέπεται κάποια συνεδρία της Επιτροπής μας εδώ μεταξύ. Η Επιτροπή, οι 40 βουλευτές, αλλά η ημερομηνία παραμένει Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε χρόνο να συνεδριάσουμε. Άλλο πράγμα είναι κάθε βουλευτή ε, να μπορεί να καταθέσει τροπολογία. Εγώ το καταλαβαίνω. Κάθε βουλευτή μέχρι τι 4 ή 3 Σεπτεμβρίου μπορεί να παρουσιάσει τι τροπολογίε που επιθυμεί και στι 4 που θα συνεδριάσουμε και θα την υποβάλουμε ω επιτροπή στο σύνολό μα. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Για να δούμε τι μα λένε οι τεχνικές υπηρεσίες εδώ πέρα.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 No, no, no, no, es, es, es la, la votación es el 5 de, de septiembre. We can extend the deadline for another like 20th of or 19th of July, July but, not more. Pero si el problema está, me dicen que solo... Κοιτάξτε, μπορούμε να παρατείνουμε μια-δυο εβδομάδες την προθεσμία. Κοιτάξτε εδώ μου λένε ότι η Κομισιόν, η 40, η Επιτροπή, ή 40 βουλευτέ μπορούν να υποβάλουν τροπολογία μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου. Έτσι έχω εδώ μπροστά στα χαρτιά. Oh, ah, Στο... Μιλάμε τότε για την Επιτροπή Προπολογισμών. Nuestro voto es el 5 de septiembre. Claro, vamos a ver. Nuestro, el voto, el voto en... Λοιπόν, εμείς στην Επιτροπή Αλληλείας θα ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Άρα θα πρέπει πριν από την 5 Σεπτεμβρίου να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες. Και η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να προετοιμαστούν όλα αυτά για να ψηφίσουμε στις 5, ποια είναι. Δεν αλλάζουν τα πράγματα αν δεν έχουμε τα στοιχεία, αν δεν έχουμε τα ποσά, δεν μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίε έτσι κι αλλιώ. Πρέπει να έχουμε τα πληροφορίες από το Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τις προτεραιότητες του, αλλά δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ε, παρουσίαση τροπολογιών ε, χωρίς να έχουμε τα σαφή αριθμητικά στοιχεία. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε ποσά για να μπορούμε να ξέρουμε, να κρίνουμε βάσει των ποσών αυτών τι μπορούμε να υποβάλουμε ως τροπολογία. Pero vamos ver, con independencia que la culpa es verdad, no δείτε, δεν φταίμε εμεί ούτε γραμματεία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μα ζητήσει να καταθέσουμε τροπολογίε επί ενός θέματος που δεν γνωρίζουμε. Από τεχνική σκοπιάς, εάν ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Αλία τις τροπολογίες, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε προθεσμία, ξέρω εγώ, Σεπτεμβρίου. Πόσο χρόνο πρέπει πριν πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες από τους συναδέλφους. Pero Ιουλίου θα λάβουμε τα στοιχεία από το Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι. Vamos a ver. Parece que en el Consejo se που ότι φαίνεται 20, τη βδομάδα 22 με 26 Ιουλίου θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Άρα τότε εμείς θα βάλουμε μια προθεσμία ε, για μας τέλη Ιουλίου για την κατασταση τροπολογιών. 29-30 Ιουλίου. Είναι ε, μοναδικός τρόπος ε, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. μήπως θα μπορούσαμε να αναβάλουμε κάπως την ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Την καθυστερήσουμε. Ε, Το πρόβλημα είναι ότι η προθεσμία αφορά τις προτάσεις που θα υποβάλουμε από τον προπολογισμό. Δεν είναι πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα του προϋπολογισμού της Επιτροπής Προεπιλογισμού που θα πρέπει να λάβει τις τροπολογίες πριν από την συνεδρίαση της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη μεταφράση τον Αύγουστο. Ο εισηγητής θα ήθελε να μας πει. Εάν ο εισηγητής ε, θεωρεί ότι δεν μπορεί να δουλέψει εφόσον δεν έχει τα στοιχεία του Συμβουλίου, δεν έχει τα ποσά, δεν αφορά το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς τους απλούς βουλευτές αλλά και τον εισηγητή. Θα πρέπει να υποβάλει το νομοδότησή του με βάση τα στοιχεία του Συμβουλίου Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να το κάνει τόσο έγκαιρα και να γνωρίσει τι θα γίνει με τα συνδύες του Συμβουλίου, θα μυρίσει τα νύχια του δηλαδή και θα βάλει τα ποσά. Ο εισηγητής θα έχει πρόβλημα. Επιτροπή Αλίας, τι, τι, σε τι θα καταθέσει τροπολογίες. Ριβελίνη, πρόεδρε, είναι σημαντικό το ζήτημα διότι κάποιοι πονηροί και δεν είμαι μεταξύ αυτών, μπορεί να πιστέψει ότι αυτές οι τόσο κοντινές ημερομηνίε κατά ε, διάρκεια των διακοπών ε, σημαίνει πως δεν επιθυμούμε να υπάρξουν τροπολογίες για κάποιες περικοπές και εγώ ως εισηγητής δεν θέλω να λάβω την ευθύνη ευχαριστώ την κυρία Φράγκα, δηλαδή να βρεθώ σε μια κατάσταση που να μην είμαι σε θέση να καταθέσω μια σοβαρή έκθεση, αλλά και να μην ε, την χάνω της στήριξης των συναδέλφων που μέσω κάποιες τροπολογίες μπορούν να αφισβητήσουν ε, κάποια ποσά τα οποία ζημιώνουν την αλία. Διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι αυτές οι ημερομηνίες ε, ε, τέθησαν τεχνιέντος ε, προκειμένου να μην μπορέσουμε εμείς να εκπληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο μας. Bien. puede hacer es... Eh, Κοιτάξτε, 31 Ιουλίου εντάξει θα είναι περίπλοκο για τη γραμματεία αλλά και για όλους μας, αλλά πιο περίπλοκο θα είναι για τους βουλευτές να δουλέψουν δίχως τα στοιχεία. Λοιπόν, 31 Ιουλίου ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών, καταληκτική. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο, είναι ό,τι θέλετε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μήπως έχετε κάποια ιδέα, μας φωτίσετε. Δεν έχω κανένα μαγικό ραβδάκι. Ριβελίνιο. Θα πρέπει να μεταθέσουμε την ημερομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου, διότι εγώ ως συγητής θα διαμαρτυρηθώ, διότι αναγκάζω τους συναδέλφους να μην καταθέσουν τροπολογίε και να μην συμφωνήσουν πάνω σε μια γραμμή του προπολογισμού, την τόσο σημαντική. Εγώ δεν μπορώ να λάβω αυτή την ευθύνη και έτσι θα πρέπει να εξεύρουμε λύση για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε με τρόπο σαφή, ξεκάθαρο, σαφή την, ε, το έργο μας. Δεν μπορούμε στις... Ε, δεν μπορούμε τώρα να μεταθέσουμε την ημερομηνία 29-30 Ιουλίου, ενώ το Συμβούλιο θα αποφασίσει 4-5 μέρες πριν. Νομίζω ότι εδώ έχουμε επικάλυψη ημερομηνιών ε, ας μεταθέσουμε την 5η Σεπτεμβρίου. Τι να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε λύση τηρώντας τον κανονισμό, αλλά είναι και, να είναι και μία λύση κατανοητή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Πέντε Σεπτεμβρίου πρέπει να συνεδριάσουμε. Εκτός αν θέλετε να μην ε, παρουσιάζουμε την γνωμοδότηση, την έκθεση. Τι θα γίνει, δεν θα έχουμε καλυθέσει τροπολογίε στην ε, εκθεσή μας. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η καλύτερη λύση. Άλλη λύση είναι να επιταχύνουμε, να πατήσουμε γκάζι και να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δεν είναι ημερομηνίε βολικές, αλλά τι να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και κάποια συνάντηση. Αλλά δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς να ξέρουμε στα τυφλά. Λοιπόν, ή στις 5 Σεπτεμβρίου δεν θα έχουμε κάποια α, θέση αποκρισταλωμένη ή θα τα ε, αναβάλουμε. Ε, αλλά εγώ 31 Ιουλίου είναι η μοναδική ημερομηνία που βλέπω. Μου είπαν ότι και πέρυσι το ίδιο συνέβη. Ότι κατέθηκαν τροπολογίες χωρίς να έχουν την ε, έκθεση του Συμβουλίου, χωρίς την απόφαση Συμβουλίου. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Εν πάση περιπτώσει. Κύριος Ριβελίνη, πρόεδρε, εσείς λέτε ότι είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, άρα πρέπει να υπάρχει πονηριά στην υπόθεση αυτή. Είναι θελημένο. Διότι το να σφάλει κανείς είναι ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Αλλά το να επιμένει και να εμένει στο σφάλμα σημαίνει ότι ε, έχει μπει ο διάβολος μέσα. Κοιτάξτε, ή παρουσιάζουμε τροπολογίες ή δεν καταθέτουμε. Τώρα, να υποβάλουμε μια έκθεση χωρίς τροπολογίες δεν έχει νόημα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίε ε, που συνεδριάζει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Άρα τροπολογιε η ημερομηνία αμετακίνητη. Μέχρι τότε μπορούμε να υποβαλουμε μια εκθεση ημερομηνία δεν εχει νοημα δεν μπορουμε να αλλαξουμε τι ημερομηνιε που συνεδριαζει η επιτροπη προπολογισμων αρα 5 σεπτεμβριου ειναι η ημερομηνια αμετακινητη μεχρι τοτε μπορουμε να κανουμε και να πούμε ότι θέλουμε. 5 όμω πρέπει να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε με τι τροπολογίε ε, στα χέρια μπορεί να υποβληθεί μία τροπολογία η οποία να λέει ότι θέλουμε, μόλον όλοι δεν γνωρίζουμε τα ποσά, ο προπολογισμό να αυξηθεί κατά τόσο. Να λάβουμε υπόψη τον... Κοιτάξτε, αυτή την τροπολογία μπορεί να την καταθέσει σήμερα όποτε θες. Αλλά δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τροπολογίες ε, χωρίς κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο εμεί παραπονιόμαστε, εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, μας βάζουν επί τελεσμένου γεγονότος, χωρίς να ξέρουμε τα ποσά. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Το ζήτημα είναι σαφές και επειδή έχουμε και άλλο θέμα θα πρέπει να προχωρήσουμε Έχουμε τον κύριο Σάντζος Πρεσέδο, κυρία Λόγαν και μετά να δούμε πώς θα κλείσουμε γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Η Ισαβέλα, έχει το λόγο. Αν κατάλαβα καλά, 5 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή. Αν θέλουμε να καταθέσουμε τροπολογίες για να αλλάξουμε τα ποσά, αυτά είναι νούμερα, αριθμοί, δεν χρειάζονται μετάφραση αυτά, Οπότε μπορούμε να κάνουμε προφορικές τροπολογίες στην Επιτροπή, αν, θα, αν το δέχεστε αυτό, για να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Pero no entendido, es decir, hasta qué momento podríamos presentar... Μέχρι πότε όμως μπορούμε να καθίσουμε τις τροπολογίες, κυρία Λεβίν. Πότε. Table them Οποτεδήποτε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Γιατί αν δεχτείτε όλοι ότι θα ε, γίνουν αποδεκτές ως προφορικές τροπολογίες, ε, όποτε θέλουμε τις ε, καταθέτουμε. If we have a agreement... Αρκεί να υπάρξει πολιτική συμφωνία, να, γίνουν, να τις αποδεχτούμε. Περίπλοκο το ζήτημα, διότι δεν γνωρίζουμε εάν όλοι θα το αποδεχθούν ή το χέρι θα πούνε αφισβητούμε τη διαδικασία αυτή. Εγώ δεν μπορώ να δεσμευθώ για τίποτα προς το παρόν. Η πολιτική συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εγκριθεί. οσδήποτε βουλευτής είναι εύκολο και ελεύθερος να αποφασίσει ότι εγώ δεν το δέχομαι. Αύριο θα δούμε έχουμε στη χειρότερη περίπτωση την 21η Ιουλίου. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον δεν θα, δεν θα κλείσει το ζήτημα αύριο. Δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Μία τελευταία πρόταση. Τουλάχιστον να μπορούμε να παρουσιάσουμε μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου μεμονωμένα ε, μία τροπολογία ή να μην χρειάζονται δηλαδή 40 βουλευτές. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό εφόσον ε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την ημερομηνία. Τουλάχιστον να μπορούμε μεμονωμένα, ε, τέλο πάντων μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, κάποιες ημέρες πριν την ψηφοφορία, να έχουμε λίγο χρόνο να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία του Συμβουλίου, τουλάχιστον να μην χρειάζονται 40 βουλευτέ. Αν υπάρχει νομική, νομικό κόλλημα, να μας το πούνε η ε, νομική υπηρεσία. Λοιπόν, στις, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου μπορούν να ε, καταθέσουν 40 βουλευτές ε, και ένα, ένας βουλευτής όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ένας βουλευτής δεν μπορεί να καταθέσει μια τροπολογία ενώ πρέπει να ε, την καταθέσουν 40. Μα εδώ η διαδικασία του προπλεσμού είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι πιστεύουμε. Το ζήτημα φέτο είναι ότι η αναγνώση του Συμβουλίου θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Εν άλλε χρονιέ γινόταν στα μέσα Ιουλίου και είχαμε 15 μέρε τον Ιούλιο να το προετοιμάσουμε. Τώρα, η, η 25η Ιουλίου είναι η ημερομηνία που θα πρέπει να ανταχθούν οι τροπολογίε που θα στηριχθούν ενδεχομένω από 40 βουλευτέ. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, να έχετε δίκιο. 31 Ιουλίου λοιπόν για την ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Καταληκτική εντάξει. Σε πολλούς δεν θα αρέσει αλλά είναι λιγότερο κακή επιλογή. Περνάμε στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως, συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών για την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταλλαγή Απόψεων επί των τροπολογιών που κατατεθεί. Κύριε Σάντσες, εδώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μια ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών που ε, υποβλήθηκαν στο σχέδιο γνωμοδότησης. Είχα την ευκαιρία να τις σχολιάσω στην Επιτροπή μας. Εννέα τροπολογίες κατέφυγαν. Του καναψί μου είναι συμβατές με το κείμενο που σας έχω υποβάλει. Αυτές, από τις εννέα τροπολογίες έξι αφορούν σε νέα άρθρα και οι τρεις προσπαθούν να συμπεριλάβουν κάποια συρωματικά στοιχεία στις ε, προτάσεις και ε, τις, έχω, τις οποίες έχω εκφράσει. Υπάρχει η τροπολογία της κυρίας Τόμας ε, για την λειτουργική οργάνωση των επιτροπών στο πλαίσιο των γραμματιών και την οργάνωση ενός συστήματος για την παρακολούθηση αυτών των ζητημάτων κάνει κάτι ερωτήσει πιο σαφής, Η κυρία Πατράου Νέβος ε, ζητάει κάποια συμπληρωματικά στοιχεία να συμπεριληφθούν στις προτάσει μου. και αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αλληλευτικής πολιτικής, κοινής αλληλευτικής πολιτικής υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για την ε, ε, μετά από τη στήγη της Λισαβόνας και αυτό δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να εκχωρήσει η Επιτροπή στον εαυτό της πρόσθετες αρμοδιότητες. Νομίζω πως αυτές οι προτάσεις είναι απόλυτα συμβατές με τις δικές μου. Υπάρχουν τώρα ακόμα έξι τροπολογίες που είναι καινούργιες, είναι νέες, που τις βλέπω με καλό μάτι, αλλά θα ήθελα να να σχολιάσουν οι καταθέτες και εγώ να κάνω μετά τα δικά μου σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αντολίν ε, Σάντσες Πρεσέτο για την έκθεσή του, ε, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Η πρώτη τροπολογία, η τροπολογία 1 νομίζω, που πρότεινα εγώ, ουσιαστικά απλώς ε, τονίζει ή συμπληρώνει ε, αυτό που έχει προβλεφθεί, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θεωρητικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα ελέγχου για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις όμως δεν υπάρχει πραγματική διαδικασία ελέγχου και αυτό αυτή ε, η εξουσία ελέγχου μοιάζει με αυτό που έγινε στον προϋπολογισμό. Ε, δηλαδή τίποτα ουσιαστικά, κοροϊδία. Γι' αυτό εκτός από αυτό που προτείνει ο εισηγητής, προτείνω να υπάρχει κάποιο είδους υποχρέωση στην ε, οργάνωση ε, της γραμματείας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και τακτική παρακολούθηση των καταξιοδότηση πράξης, κάτι το οποίο πρέπει να εγγράφεται τακτικά στην ημερήσια διάταξη. Ξέρω εγώ ε, σε μία-δύο συνεδριάσεις Επιτροπής ε, κατέτος και να γίνεται εξέταση της παρακολούθησης ε, των καταξιοδότηση πράξεων. Για την τροπολογία 2, το σημείο αφετηρίας είναι πάνω κάτω το ίδιο. Συγγνώμη, μιλάτε και δεν ακούω. Έλεγα λοιπόν, ε, πάλι ξεκινώντας από την ιδέα ότι το Κοινοβούλιο έχει τον, την εξουσία του ελέγχου, αλλά αντί να το κάνει εκ των προτέρων, ε, διευκρινίζοντας εκ των προτέρων τα κριτήρια για τα βάση των οποίων δεν θα διαφωνήσει με αυτές τις κατεξοδότηση πράξεις, εξασφαλίζουμε ε, προτεραιότητα ε, για το Κοινοβούλιο ε, σε σχέση με αυτό που θα εγκριθεί ή που δεν θα εγκριθεί στη συνέχεια από το Κοινοβούλιο. Και τρίτη τροπολογία, πάλι η ίδια ιδέα του ελέγχου από το Κοινοβούλιο, γιατί είναι ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου, και για να υλοποιηθεί όντως αυτός ο ρόλος με αποτελεσματικό τρόπο, η δημοσίευση των πράξεων αυτών να είναι πιο διαφανής να υπάρξει οργάνωση της ε, διάδοσης αυτών των πράξεων, ε, να είναι λιγότερο ε, κρυμμένη από ό,τι γίνεται από τη σχή σήμερα με ένα εργαλείο πληροφορικής, όπως μια βάση δεδομένων για παράδειγμα, κάποιου είδους ε, κατάλογος, κατάλογος ανακατηγορία κατεξιοδότηση πράξης, που θα δίνει τη δυνατότητα να ε, γίνεται καλύτερος δημοκρατικός έλεγχος από πλευράς Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τροπολογίες ε, που ουσιαστικά μεταγράφουν ε, τις, τους προσανατολισμούς του εισηγητή, πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον έλεγχο, η εξουσία του, του οποίου δόθηκε από τον νομοθέτη στο Κοινοβούλιο και μιλάω για τη συνθήκη της Λισαβόνας και που δεν ε, έχει σήμερα το Κοινοβούλιο ε, ουσιαστικά κανένα μέσο για να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο. Κάνα σχόλιο, Κομισιόν, κύριος Πρεζέδο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση των τροπολογιών από την κυρία Τόμα. Συμφωνώ με τις θέσεις της Σημασία έχει το Κοινοβούλιο να καθορίσει τις, ε, τα κριτήρια και τα της πράξης είναι αυτές οι οποίες προσδιορίζονται κατά περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κάποια κριτήρια και υπάρχουν και κριτήρια σκοπιμότητας στο κάτω-κάτω. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι περιστάσεις ε, και θα μπορούσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε μια σειρά κριτηρίων που θα δίνουν συνέπεια και συνεκτικότητα στις ε, θέσεις μας και στις προτάσεις μας. Επίσης θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το οποίο θίγει ότι υπάρχει δυνατότητα για ύπαρξη μια βάση δεδομένων στην οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να γνωρίζουμε το θέμα των ευθυνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ως εκ τούτου λοιπόν δεν έχω καμία δυσκολία να τις στηρίξω αυτές τις ε, προτάσεις της κυρίας ε, Τόμας. Ε, οι κατεξιώσεις πράξεις δεν έχουν κάποιο χρονικό όριο εν το οποίο ισχύουν και ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται για κάποιος χρονικός περιορισμός. Υπάρχουν τρεις προτάσεις λοιπόν που έχει παρουσιάσει και ο κύριος Γκάλαχερ. Από τις τρεις αυτές προτάσεις ε, συμφωνώ. Μπορώ να συμφωνήσω με την ε, μικροδιαχείριση που όπως αναφέρεται. Έχουμε όμως ε, μια νομοθεσία η οποία είναι περίπλοκη και η διαδικασία της συναπόφασης είναι κάτι το σχετικά άκαμπτο και οδηγεί σε καθυστερήσει ε, Τώρα δεν, σύμφω, δεν ξέρω αν πρόκειται για ζήτημα μετάφραση. Ε, δεν έχω το αγγλικό κείμενο, μιλάει για εκτελεστικέ αρμοδιότητες. Ε, Οι πράξεις δεν είναι εκτελεστικές και δεν μπορούν να εκχωρηθούν. Ο απλά δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να υποβάλλονται αυτέ οι πράξει. Εντάξει, είναι τεχνικής φύσης συζήτηση, στο συμφωνώ με την ε, αποφυγή της ε, μικροδιαχείριση ε, και επίση θεωρώ σημαντικό και το τονίζει εδώ η τροπολογία τη στήριξη στη γραμμή που είχε αποφασίσει η η σύσκεψη των Προέδρων νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση που αναφέρει την έλλειψη αξιοπιστίας όταν τελικά οδηγούμεθα σε κάποιες ε, πολιτικές ε, που δεν μπορούν να θεσπιστούν διότι τα δύο θεσμικά όργανα δυνατούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει κάποια μνήμη αυτών των προβλημάτων και το τελικό κείμενο θα ανθρωποποιηθεί καταλήλως. Συμφωνώ λοιπόν με αυτές τις ε, τροπολογίες, διότι συμπληρώνουν τις προτάσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, ε, θεωρούμε ότι τελείωσε η σημερινή μας συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους Γερμανείς και οι Γερμανείς ευχαριστούν τον Πρόεδρο. Θα τα πούμε αύριο.